Buenos Καλημέρα σα. Θα ξεκινήσουμε. Θα κάνω μια πολύ σύνταμη εισαγωγή. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ε, μέρα. Ε, βέβαια η χθεσινή νύχτα ήταν πολύ μεγάλη. Ε, συζητούσαμε μέχρι τις 4 παρατέταρτο το πρωί τα θέματα του τριμερούς διαλόγου, αλλά θα ήθελα να πω ότι καλώς κάναμε γιατί καταλήξαμε σε μια πολύ σημαντική συμφωνία και πάντα όλοι κάτι παραχωρούμε για να κερδίσουμε όλοι πολλά και τελικώς αυτό κάναμε και σε αυτή την περίπτωση. Χρειάστηκε να ε, ε, παραχωρήσουμε κάποια πράγματα, αλλά ε, για πρώτη φορά αποφασίστηκε η πρώτη μεταρρύθμιση σε συναπόφαση. Ε, και επομένω έχει μια ισχύ την οποία δεν είχε μέχρι τώρα και είναι ε, μια διαδικασία η οποία δεν ήταν εύκολη, είχε πολλές συζητήσεις, πολλές συνεδριάσεις, πολλές ε, διαπραγματεύσεις, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι καταλήξαμε σε συμφωνία. Σήμερα λοιπόν είναι ωραία μέρα. Και μάλιστα, εάν ε, το συνδυάσουμε και με μία κρόαση για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που είναι ε, βιώσιμη ευκαιρία για την αλία και την υδατοκαλλιέργεια, ακόμα περισσότερο, διότι ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Έχουμε σήμερα ένα πολύ φιλόδοξο και πλήρες πρόγραμμα και θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω όλους όσους συμμετέχω, τους προσκεκλημένους μας άτομα εγνωσμένου κύρους. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή μια πρόταση οδηγίας για τον καθορισμό ενός πλαισίου για τον ολοκληρωμένο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και η βασική ιδέα αυτής της οδηγίας ήταν να διασφαλίσει ότι η αύξηση των θαλάσσιων πόρων και η χρήση των διαφόρων δυνατοτήτων που μας προσφέρει η θάλασσα θα είναι υποφελής για όλους. Το θέμα βέβαια ε, είναι πάρα πολύ ευρύ και η Επιτροπή Αλίας, ε, όπως και πρέπει να κάνει, ενδιαφέρεται κυρίως για την ε, βιωσιμότητα της αλίας και της υδατοκαλλιέργειας και αυτό είναι και το επίκεντρο της σημερινής μας ακρόασης. Αλλά θα αναλύσουμε και διάφορα ε, σημαντικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους, τα θέματα του σχεδιασμού και τα συμφέροντα διαφόρων τομέων και κλάδων Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ακρόαση και ελπίζω στο επόμενο διάστημα να μπορέσουμε να δούμε πώς ε, θα προχωρήσουν όλα αυτά τα θέματα που έχουν ξεκινήσει. Ε, θα έχετε δει το πρόγραμμα της ακρόασης φαντάζομαι. Ε, ε είναι καταμερισμένο σε τρία πάνελ διάρκειας μίας ώρας το καθένα και αυτό το οποίο θα ήθελα ευθύ εξ αρχής είναι οι ομιλητές να προσπαθήσουν να τηρήσουν τα χρονικά όρια για να είναι μια δυναμική η στη σημερινή και να μπορέσουμε να έχουμε και χρόνο για συζήτηση που πάντα είναι σημαντική. Πριν δώσω το λόγο στην πρώτη συγγήτρια, η οποία θα ε, κάνει και την αρχική εισαγωγή, την ε, κυρία Ιζαμπέλ Τομάς, θα πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη, διότι οι χθεσινές συνέπειες έρχονται σήμερα. Ε, πρέπει να συναντηθούμε με την Επίτροπο, τον ε, Υπουργό Κόβενε και την Ισηγήτρια για να κάνουμε μια συνέντευξη τύπου ε, διάρκειας μιας ώρας. Ε, βέβαια με εκπροσωπεί επάξια ο Αντιπρόεδρος, ο κύριος Στίβενσον, ο οποίος ε, σήμερα θα προεδρεύσει. Ευχαριστώ πολύ σε όλους και για να ξεκινήσουμε με το πρώτο πάνελ να δώσω το λόγο στη συνάδελφο την Ιζαμπέλ Τομάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα καταρχάς ε, να συγχαρώ τη διαπραγματευτική ομάδα για την συμφωνία στην οποία καταλήξαμε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ευχαριστίες. Καταρχάς προς τους συναδέλφους, ε, παρά το γεγονός ότι σήμερα δεν είναι και πολλοί συνάδελφοι λόγω της κατάστασης, να ευχαριστήσω και τους ομιλητές που δέχτηκαν να έρθουν και να μας παρουσιάσουν τις απόψεις τους για την ακρόαση αυτή και να ευχαριστήσω ιδιαίτερως και την ομάδα των φιλελευθέρων που ανέλαβε την πρωτοβουλία για αυτή την ακρόαση και ε, διευκόλυνε ιδιαίτερα ε, στην ε, ε, κατάρτιση της σύνθεσης των ομιλητών στα διάφορα πάνελ. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την πρωτοβουλία, για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και πιο συγκεκριμένα το θαλάσσιο χωροτεξικό σχεδιασμό που κατά την άποψή μου είναι τα βασικά στοιχεία της γαλάζιας βίβλου. Ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι το μέσο, να μην ξεχνάμε, γιατί ο στόχος είναι η ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων εργασίας, και φυσικά ελπίζουμε ότι θα δημιουργήσουμε επιπλέον 1,6 εκατομμύριο θέσεις εργασίας ε, ε, με τις νέες ε, δραστηριότητες που θα υπάρχουν στη θάλασσα και θέλουμε να έχουμε φυσικά και ανάπτυξη από σήμερα μέχρι το 2020. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα αναπτυχθούν εκ νέου οι δραστηριότητες αυτές και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να έχουμε και τα κατάλληλα μέσα για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Ε, μόλις είπε και ο κύριος Πρόεδρος, για να επιτύχουμε το στόχο αυτό θα πρέπει να αποφύγουμε δύο παγίδες. Η πρώτη παγίδα θα είναι να, ξανά, επανα, να επαναλάβουμε τα σφάλματα του παρελθόντων, δηλαδή την κατασπατάληση των φυσικών πόρων και την ε, βάθμιση του περιβάλλοντος. Και δεύτερον, να μην επιτρέψουμε οποιαδήποτε ανάπτυξη επειδή υπάρχουν ε, κάποιες ε, υπερβολικές απαιτήσει σε κάποιες περιπτώσεις διότι λαμβάνονται μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που θα είναι ίσως και υπερβολικά ή θα είναι ακραία διότι τα μέτρα προστασίας κάποιων συμφερόντων μπορεί να αποτρέψουν την ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε να πέσουμε σε αυτές τις δύο παγίδες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε βιώσιμη και εφόρο ανάπτυξη και ε, ο θαλάσσιος χωροτεξικό σχεδιασμός ε, θεωρώ ότι μας επιτρέπει να αναζητήσουμε τη δέουσα ισορροπία μεταξύ ε, των διαφόρων συμφερόντων αφενός και της προστασίας του περιβάλλοντος αφετέρου, αλλά θα πρέπει να βρούμε και τη δέουσα ισορροπία μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων και να βρούμε και την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των πολυτομιακών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα η Αλία, και των μελλοντικών δραστηριοτήτων διαθέτουμε ήδη πριν ξεκινήσουν αυτές οι μελλοντικές δραστηριότητες ε, ε ισχυρές ε, πιέσεις ε, στις παράκτιες περιοχές. Είναι πολλές οι δραστηριότητες, η αλληλεία, η καλλιέργεια και άλλες και αν αυξηθούν φυσικά οι χρήσεις του θαλάσσιου χώρου θα αυξηθούν και οι πιέσεις. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι Θεωρώ ότι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνούμε για το ε, κατά πόσον είναι κατάλληλα τα μέτρα τα οποία προτείνονται για τη διαχείριση των ακτών για διάφορους λόγους. Καταρχάς, διότι η θάλασσα και οι παράκτιες περιοχές ε, παρά το γεγονός ότι θεωρούνται, ότι θεωρούνται ξεχωριστά ε, πράγματα, επειδή υπάρχει αυτή η στοιχή στη μέση, η ακτή στη μέση, στην πραγματικότητα είναι κοινέ οι δραστηριότητες και η ζωή στις παράκτιες περιοχές και στη θάλασσα ε, είναι αλληλένδετη. Οι πιέσει είναι μεταξύ τους ε, πολύ σημαντικές. Και το δεύτερο είναι ότι είναι πολλοί οι παράγοντες που συμμετέχουν ε, ε, στην διαχείριση και επομένως θα πρέπει να οργανωθεί αυτή η ολοκληρωμένη διαχείριση κατά τρόπον, ε, και εδώ θα προσθέσω και ένα τρίτο στοιχείο, ώστε να συμπεριλάβει όλα τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά στοιχεία, και ε, το γεγονός ότι είναι πολλαπλά τα ενδιαφέροντα. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο στοιχεία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω και ένα τρίτο τώρα. Το τρίτο είναι η συζήτηση για το κατά πόσο είναι ενδιαφέρουσα αυτή η οδηγία. Νομίζω ότι ε, είναι από τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν περισσότερο. Ε, είναι κάτι το οποίο συζητάται σε πολλά κράτη-μέλη, διότι πολλά κράτη-μέλη ήταν είτε επιφυλακτικά είτε αντίθετα, διότι δεν θέλουν ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός να οργανωθεί από μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από πλευράς μου, παρά το γεγονός ότι θα ακούσουμε και τι έχουν να πούν οι ομιλητές, θεωρώ ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός έχει κάποιο ενδιαφέρον, διότι καταρχάς μιλάμε για τη θάλασσα. Ε, και η θάλασσα έχει πολύ πιο σημαντικές ε, πτυχές σε διασυνοριακό επίπεδο από ότι στο, ε, στη γη, στην ξηρά. Ε, και ακόμα και η αναψυχή, ο τουρισμός περιλαμβάνουν ένα στοιχείο κίνησης και είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχουν κανόνες που θα είναι διαμέτρου αντίθετοι από τη μία χώρα στην άλλη. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω ότι συνεχώς, ακόμα και εδώ στην Επιτροπή μας, επισημαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε κοινά κριτήρια, κοινού κανόνες, κοινέ μεθόδους, ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε το τι συμβαίνει στη θάλασσα. Και αυτό, κατά την άποψή μας, θα επιτρέψει, ή τουλάχιστον αυτό είναι ένας από τους στόχους που θέτουμε, είναι να μπορούμε να μιλούμε για το ίδιο πράγμα με τα ίδια μέτρα και τις ίδιες μεθόδους. Δεν θα ήθελα εδώ να καθυστερήσω περαιτέρω ε, την Επιτροπή. Ε, ξέρω τι γίνεται με τις ακροάσεις. Θα ήθελα λοιπόν ε, ως πρώτο συμπέρασμα, και δεν τολμώ καν να πω τον όρο συμπέρασμα, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε τις οικονομικές και κοινωνικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες και θα πρέπει προς το συμφέρον όλων μας να προσπαθήσουμε να ε, υλοποιήσουμε αυτό το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό για να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και θέσεις εργασίες και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τίνουμε βίκονους και εμείς αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ακούσουμε και όλες τις απόψεις ε, και όλες τις διαφορετικές εμπειρίες ώστε να εξεύρουμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ημών αλλά και μεταξύ οικονομικών συμφερόντων και προστασίας ε, του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του παράκτιου περιβάλλοντος και επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν και κάποιες δραστηριότητες και χρήσεις που μπορεί να φαίνεται ότι είναι αντίθετες η μία προς την άλλη και θα πρέπει σε αυτή τη διαχείριση ε, να πούμε ότι όντως υπάρχουν και κάποιες εξουσίες ε, οι οποίες θα μπορούσαν και αυτές να είναι αντίθετες η μία με την άλλη. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου πάντα την ε, ανάπτυξη της θάλασσας και πριν ολοκληρώσω πρέπει να παρουσιάσω και τους δύο πυρογνώμονές μας που θα παρέμβουν τώρα. <coughs> <laughs> Donc, euh, Καταρχάς, η κυρία Κάρλα Μοντέζη από την ε, Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ και στη συνέχεια ο κύριος Αρμάν Κεντέλ, μέλος της Εθνικής Επιτροπής ε, Αλίας ε, στην Γαλλία. Ευχαριστώ και τους δύο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Ιζαμπέλ Τομάς είναι κρίμα που δεν είναι <clears throat> περισσότεροι ευρωβουλευτέ παρόντες, ε, αλλά όπως ακούσατε ε, τον πρόεδρο να λέει, η συζήτηση συνεχίστηκε μέχρι τις 4 ώρα το πρωί, αλλά λόγω του ενδιαφέροντος του τύπου οι περισσότεροι δεν κοιμήθηκαν πριν τις 6.30 το πρωί. Δεν περιμένω λοιπόν ε, να δω ε, τόσο πρωί του ε, συναδέλφους και λυπάμαι γι' αυτό, διότι ε, αν ήταν παρόντες θα είχαν ακούσει μια εξαιρετική παρουσίαση της κυρίας Τομάς. Να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Κάρλα Μοντέζη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Τομάς για την επισκόπησή της. Να σα συγχαρώ και για τις χθεσινοβραδινέ διαπραγματεύσει που αποτελούν πολύ σημαντικό βήμα. Σας ευχαριστώ και την πρόσκληση αυτή να παρουσιάσω την ε, πρόταση της ε, Κομισιόν. Είναι επίκαιρη η ακρόαση αυτή που θα μας επιτρέψει να συζητήσουμε τη σημαντική αυτή πρόταση. Όπως ξέρετε, τον τελευταίο χρόνο η Κομισιόν έχει αναλάβει σημαντική πρωτοβουλία για προώθηση της ε, βιώσιμης ανάπτυξης της θαλάσσιας και της παράκτιας οικονομίας. Πρόκειται για τη λεγόμενη γαλάζια ανάπτυξη και πιστεύουμε ότι για να συμβάλλουμε ε, στην επίτευξη της στρατηγικής Ευρώπη 2020 έχουμε εντοπίσει πέντε τομείς θαλάσσιους όπου πιστεύουμε ότι μπορεί να έχουμε ανάπτυξη. Και όταν μιλάμε για ανάπτυξη μιλάμε για θέσεις απασχόλησης. Έχουμε εντοπίσει λοιπόν αυτούς τους πέντε τομείς, κάποια σημεία συμφώνησης ε, και ε, πιθανές ε, πολιτικές παρεμβάσεις. Όλα τα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται σε μια στρατηγική η οποία εγκρίθηκε πέρσι σε υπουργική διάσκεψη στην Λεμεσό. Είναι η λεγόμενη διακήρυξη της Λεμεσού. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελεί στοιχείο κλειδί της στρατηγικής αυτής. Πρόκειται για μέσο το οποίο θα μας επιτρέψει να προωθήσουμε την θαλάσσια ανάπτυξη, διευκολύνοντας ε, την ανάπτυξη ε, τομέων σε ένα πλαίσιο αυξανόμενου ανταγωνισμού όσον αφορά το χώρο. Και βλέπετε τα στοιχεία, τα νούμερα που ε, δείχνουν το πρόβλημα. Ας επικεντρωθώ σε ένα παράδειγμα. Την ηχθειοκαλλιέργεια ήταν ένας από τους πέντε τομείς που εντοπίστηκαν ε, και όπου υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης. Ε, έχουμε υιοθετήσει στρατηγικέ κατευθυντήριες γραμμέ για τον τομέα τη ηχθειοκαλλιέργεια ε, και μπορούμε να πούμε ότι η εξαιρετική ποιότητα των θαλασσινών τη Ευρώπη θα πρέπει να συμβάλλουν στη σημαντική ανάπτυξη τη αλλά βλέπουμε ότι λιμνάζει ε, η παραγωγή στην Ευρώπη σε αντίθεση με την ισχυρή ανάπτυξη που βλέπουμε σε άλλε περιοχέ. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εάν κοιτάξουμε την ε, συνολική κατανάλωση ψαριών και θαλασσινών, βλέπουμε ότι το 25% προέρχεται από αλληλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 10% από ηχθειοκαλλιέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 65% προέρχεται ε, από εισαγωγές. Ποιο είναι λοιπόν ο στόχο μας. Ο στόχο μας είναι το 65% το κενό, το, το, το κενό αυτό, ανάμεσα στην κατανάλωση και την παραγωγή να το συμπληρώσουμε. Ε, και με την παρούσα παραγωγικότητα κάθε 1% ε, αυξημένης κατανάλωσης ε, ε, ψαριών και θαλασσινών που παράγεται από την ιχθυοκαλλιέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούμε 3 με 4 χιλιάδες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θέλουμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να δημιουργήσουμε ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για την ηχθειοκαλλιέργεια και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με την ε, την ε, μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής ε, που θα δώσει το νομικό υπόβαθρο. Θα είναι όμως αυτό δυνατό μέσω του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, διότι έτσι παρέχουμε το καλύτερο εργαλείο για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον τομέα αυτών, διευκολύνοντας την πρόσβαση στο νερό για οποιοδήποτε πρόγραμμα ηχθειοκαλλιέργειας. Αυτό αποτελεί απλά ένα παράδειγμα ενός από τους πέντε τομείς όπου έχουμε που έχουμε εντοπίσει όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερες θέσει απασχόλησης. Τι είναι λοιπόν ο θαλάσσιος χωροταξικός ε, σχεδιασμός. Ε, για να είμαι σύντομη, θα ήθελα να ε, επικεντρωθώ σε κάποιους βασικούς τομείς. Πολύ σύντομα να πω ότι πρόκειται για την διοργάνωση του πού και πότε πραγματοποιούνται ανθρώπινες δραστηριότητες στη θάλασσα. Στόχος είναι να δημιουργηθούν σχέδια τα οποία να εντοπίζουν τον ε, πιο την πιο αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση του θαλασσίου χώρου. Αυτό που θέλουμε είναι μια διαφανής διαδικασία που να βασίζεται στην εμπλοκή των ε, ε, ενδιαφερόμενων ομάδων. Με τη συμμετοχή όλων των βασικών οικονομικών τομέων που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα και πρέπει να είναι πολετομεακή η προσέγγιση. Θέλουμε δηλαδή ένα εργαλείο το οποίο να είναι ουδέτερο ως προς τον τομέα ε, για, την, για τον συνδυασμό των ε, ανθρωπίνων ε, δραστηριοτήτων και διαχείριση του, της των επιπτώσεων τους στο θαλάσσιο περιβάλλον. Μιλάμε για την αλία, την ηχθειοκαλλιέργεια, ενέργεια, μεταφορές ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλες αυτές οι δραστηριότητες στη θάλασσα ε, χρειάζονται χώρο. Χρειάζονται πρόσβαση στη θάλασσα. Κατά την ε, προετοιμασία της πρότασης εντοπίσαμε τέσσερα σημαντικά προβλήματα τα οποία βλέπουμε να υπάρχουν και στου τομεί αλληλεία και ηχθειοκαλλιέργεια. Το πρώτο ήταν αυτό που μόλι ανέφερα. Ε, οι συγκρούμενε αξιώσει όσον αφορά τον ε, θαλάσσιο χώρο και την πρόσβαση στη θάλασσα. Δεύτερον, το γραφειοκρατικό άχθο. Ε, όσον αφορά την ηχθειοκαλλιέργεια, είναι σημαντικό το γραφειοκρατικό άχθο. υπολογίσαμε ότι ο χρόνος απόκτησης αδείας για αιωλικά πάρκα είναι έξι μήνες. Ε, σε κάποια κράτη-μέλη ε, η άδεια για ε, καταστάσει ηχθειοκαλλιέργεια σε κάποια κράτη-μέλη απαιτεί δύο με τρία χρόνια. Θέλουμε λοιπόν να μειώσουμε το γραφειοκρατικό άρθρο και να επιταχύνουμε τι επενδύσει. Επίσης είδαμε ότι δεν υπάρχει η βέλτιστη εκμετάλλευση των οικονομικών δυνατοτήτων. Εάν βάλουμε σε ένα ε, πολυτομεακό σχέδιο όλες τις δραστηριότητες ε, που αφορούν τη θάλασσα, θα δούμε αμέσως τα ωφέλη που μπορούμε να πετύχουμε απλά με τον καλό συνδυασμό όλων των ε, δραστηριοτήτων. Το τέταρτο πρόβλημα που μόλις αναφέρθηκε είναι η περιορισμένη διασυνοριακή συνεργασία. και στη θάλασσα είναι πιο σημαντικός ο διασυνοριακός συντονισμός ε, από ό,τι αλλού. Ε, να αναφερθώ στο οικοσύστημα, τα παιδεία αλληλείας, ε, είναι κάποια από τους τομείς όπου η διασυνοριακή συνεργασία είναι απαραίτητη. Η διαπίστωση των προβλημάτων αυτών οδήγησε την Κομισιόν να υποβάλει πρόταση τον περασμένο Μάρτιο. Ε, η πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ε, και μια ολοκληρωμένη διαχείριση των ακτών. Γιατί οδηγία, διότι η μελέτη αντικτύπου ε, έλεγε σαφέστατα ότι μια νομικά δεσμευτική προσέγγιση είναι το πιο κατάλληλο μέσο για να διασφαλίσουμε τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ωφέλη. Έτσι λοιπόν μπορούμε να έχουμε συνεργασία συνεργασία μεταξύ των κρατών ε, ε, και να σεβαστούμε ε, τα οικολογικά όρια του οικοσυστήματος. Έχουμε για παράδειγμα τη σύσταση της οδηγίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ακτών που λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε τα ωφέλη αυτά εάν δεν έχουμε ένα νομικά δεσμευτικό μέσο. Αλλά βέβαια θέλουμε να έχουμε ένα απλό δεσμευτικό μέσο. Έτσι λοιπόν στην πρόταση αυτή επιβάλλουμε λίγες υποχρεώσεις. Η πρώτη είναι να υπάρχουν σχέδια, να υπάρχει μια στρατηγική που να διευκολύνει τη συνύπαρξη και να αποτρέπει την σύγκρουση ανάμεσα σε διάφορες ε, δραστηριότητες. Ε, και με τους πολιτικούς στόχους που ήδη έχουμε ε, στην ε, ε, Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να το πετύχουμε αυτό. Θέλουμε λοιπόν όχι να ευνοήσουμε ένα τομέα, αλλά να συμπεριλάβουμε όλους τους στόχους κλειδιά που μπορούμε να έχουμε στην ενέργεια, στις μεταφορές, στην αλληλεία, όσον αφορά το περιβάλλον και όσον αφορά την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Έχουμε λοιπόν ε, μια πολιτική ε, υιοθετημένη σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατά την εφαρμογή της οδηγίας δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να προσθέσουν άλλους τομείς που θεωρούν σημαντικούς. Έχουμε λοιπόν κάποιες πολιτικές που θεσπίζονται και με την συνθήκη, αλλά και τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν ποιες είναι οι τομεακές τους προτεραιότητες. Η βασική υποχρέωση που επιβάλλει η οδηγία είναι να αναπτυχθεί ε, και να εφαρμοστεί ε, ένα ε, σχέδιο θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού ή σχέδια, δηλαδή δεν θέλουμε απαραίτητα ένα σχέδιο για όλα τα κράτη-μέλη. Σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε συντονισμό ε, μεταξύ των διαφόρων αυτών σχεδίων και στρατηγικών ε, για να διασφαλίσουμε αυτό που ανέφερε η κυρία ε, Τομάς, την σχέση στεριάς και θάλασσας. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε μία από τις δύο αυτές πτυχές. Επίσης σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και με τρίτες χώρες ε, για να διασφαλίσουμε μια συνεκτική προσέγγιση ε, σε όλες τις θαλασσίες λακάνες ε, και επίσης υπάρχει η υποχρέωση διαβούλευσης με τις ομάδες ενδιαφερομένων. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε τέτοιες υποχρεώσεις σε διαδικαστικού χαρακτήρα. Δεν ε, προσθέτουμε κάποιο νέο τομέα. Θέλουμε να αποφύγουμε ε, οποιαδήποτε επικάλυψη εργασιών. Όταν ε, λοιπόν μιλάμε για την αναλογικότητα και την επικουρικότητα, να απαντήσω σε κάποιες πιθανές ερωτήσεις. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να τονίζει ότι τα κράτη-μέλη διατηρούν την πλήρη αρμοδιότητα ε, σχετικά με το τι και πού ε, θα έχουν σχεδιασμό. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται ε, σύμφωνα με τις δομές διακυβέρνησης των κρατών μελών, τοπικές ή εθνικές. Δεν λέμε δηλαδή στα κράτη-μέλη που ή ποια αρχή θα πρέπει να ετοιμάσει τα σχέδια. Αυτό θα, αποτελεί, αυτό θα γίνεται σύμφωνα με τη δομή του κάθε κράτους μέλους. Ε, θέλουμε σαφώς να αναφέρεται ποια θα είναι η αρμόδια εθνική αρχή, διότι οι ομάδες ενδιαφερομένων ε, λένε ότι αυτό σε πολλά κράτη-μέλη είναι πρόβλημα, ότι δεν γνωρίζουν ε, ποια είναι η βασική αρχή. Ζητάμε δηλαδή από το κράτος μέλος να διορίσει αρμόδια την αρχή που θα είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και τη στρατηγική. Και κατόπιν τα κράτη-μέλη μπορούν να εργαστούν με βάση τους μηχανισμούς που έχουν και την πολιτική που έχουν. Δεν θα υπάρξουν λοιπόν νέες υποχρεώσεις για ε, τομείς που αφορούν τη θάλασσα, ούτε επικάλυψη εργασιών. και η πρόταση σέβεται απόλυτα το προνόμιο των κρατών μελών, το δικαίωμα των κρατών μελών να διαμορφώνουν ε, το περιεχόμενο των ε, σχεδίων και στρατηγικών ε, στις, στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προτεραιότητες τους, καθώς και τις εθνικές και τους εθνικούς τομεακούς πολιτικούς στόχους. Δεν θα υπάρχει λοιπόν παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το περιεχόμενο ε, των σχεδίων και στρατηγικών. Και δεν θα παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο δικαίωμα των κρατών μελών ε, για ε, χωροταξικό σχεδιασμό. Και φαντάζομαι ότι έτσι έχω ήδη απαντήσει σε ερώτηση που μπορεί να τεθεί από πλευρά των κρατών μελών. Κλείνοντας, να πω ότι ο γενικός στόχος που θέλουμε να πετύχουμε είναι να πετύχουμε περισσότερη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους βασικούς θαλάσσιους τομείς και μάλιστα όσο γίνεται πιο σύντομα. Και όταν μιλάμε για τη θάλασσα, μιλάμε φυσικά και για την αλληλεία ε, και την ηχθειοκαλλιέργεια. Ε, στόχος της πρότασής μας είναι να ε, συμβάλλει στην περισσότερη ανάπτυξη και ε, περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αλίας. Ελπίζουμε να υπάρχει ε, συμφωνία ε, ανάμεσα στα θεσμικά όργανα πριν το τέλος της θητείας. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσίαση, κυρία Μοντέζη. Ήταν ε, πολύ ενημερωτική σε ό,τι αφορά τι προτάσεις της ε, Κομισιόν και την οδηγία. Προτείνει, ειδικά για μένα. Τώρα, θα δώσω το λόγο στον κύριο Αρμό Καντέλ, μέλο της Εθνικής Επιτροπή Αλία και τη της Γαλλίας. Merci, Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ που θα ακούσετε τη φωνή της Εθνικής Επιτροπής Αλίας και Εχθιοκαλλιέργειας Γαλλίας. Θα μιλήσουμε για την διαχείριση των ε, υγρής μορφής ε, μέσων περιβαλλόντων και ιδιαίτερα ε, των θαλασσών. Μιλάω για αυτά τα περιβάλλοντα αυτά τα μέσα τα οποία ε, έχουν ιδιαιτερότητες σε σχέση ε, με τα χερσαία μέσα. Χρειάζονται λοιπόν, έχουν διαφορετικές ανάγκες ε, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ελαστικότητα. Η συμβίωση εκεί είναι σημαντική γιατί είναι χώροι όπου μοιράζονται οι δραστηριότητε, Τα αλληλευτικά, οι αλληλευτικοί πόροι είναι δυναμικής φύσεως και ακόμα και πρόσφατα στο παρελθόν χαρακτηρίζονται αυτές οι ζώνες ε, από συγκρουσιακό χαρακτήρα. Για να λυθούν οι, αυτά τα εσωτερικά προβλήματα έχουν, έχουμε συστήματα ε, συμφωνίες μεταξύ των διαφόρων ε, φορέων, συστήματα αδειοδότησης κλπ. Αλλά ε, θα πρέπει ε, να καθορίσουμε και τις σχέσεις με τους νεοαφιχθέντες της γαλάζιας οικονομίας, τους νεοαφικνιόμενους για την ακρίβεια, προκειμένου να αποφύγουμε σύγκρουση στο μέλλον. Η... Το οι, δυνατότητε οι δυνατότητες που προκύπτουν είναι τεράστιες για το μέλλον. Ο αλληλευτικός τομέας ε, παρακολουθεί πολύ προσεκτικά το χωροταξικό σχεδιασμό ε, και το σχεδιασμό των χρήσεων. Οι τεχνικές ε, έχουν διευρύνει τα όρια των δραστηριοτήτων. Δεν είναι δυνατό όμως πάντοτε να πηγαίνουν πιο μακριά και πιο βαθιά. Γι' αυτό το λόγο η χωροταξία στη θάλασσα θα πρέπει να τηρεί ένα διακλαδικό, ένα διατομεακό πρωτόκολλο με τη συνεργασία όλων. Ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι στρατηγικής ε, φύσεως και όχι μόνο γεωγραφικής. Είναι ένα εργαλείο που θα μας επιτρέψει ε, να προγραμματίσουμε στην κατάλληλη κλίμακα της χρήσης με κατάλληλη προσαρμοστικότητα ε, η οποία είναι απαραίτητη δεδομένου ότι πολλά λιευτικά αποθέματα ε, κινούνται ε, και είναι πολύ δυναμικά, επηρεάζονται και από το περιβάλλον. Θα πρέπει ο χωροταξιός ιδανός να επιτρέπει την ε, πολλαπλές χρήσεις ε, και θα πρέπει να εμπλέξει όλους τους ενδιαφερόμενους και φορείς από νωρίς, από την αρχή. Ε, ε, ήδη ο διασυνοριακός συντονισμός μεταξύ ψάρων διαφορετικών εθνικότητων υπάρχει. Θα πρέπει όμως να γίνουμε περισσότερους φορείς και όσο πιο νωρίς γίνεται στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού. Ε, η, τα αλλιεύματα ε, Ευρωπαϊκή Ένωση που καταναλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% της συνολικής κατανάλωσης και υπάρχει κίνδυνος να εξαφανιστούν, να μηδενιστούν οι αλευτικές μας ικανότητες. Ε, ταυτόχρονα ε, φύσταται ο κίνδυνος πλήρους εξάρτησης από τις εισαγωγές μας. Αυτό είναι στρατηγικό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η βιώσιμη ανάπτυξη των αλληλευτικών δυνατοτήτων μας συνδέεται στενά με τη διαχείριση ασφαλώς, αλλά όλο και περισσότερο με τις ε, εξελίξεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της, με το, ε, με το περιβαλλοντικό, την περιβαλλοντική κατάσταση και με τη μόλυνση. Οι αλληλείς αντιμετωπίζουν καθημερινά αυτές τις επιπτώσεις. Η οδηγία 56 του 2008 ε, συνδέεται άμεσα με, το, με το θέμα αυτό. Ε, αυτή η, η περιβαλλοντική πτυχή θα πρέπει να συμπληρωθεί με ε, μια απέτηση κοινωνικής αποδοχής των εισαγωγών. Αυτό είναι απαραίτητο διότι οι εισαγωγές δεν θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν ε, να αντιπροσωπεύουν την εξαγωγή μιζέριας προς τις ε, χώρες από τις οποίες εισάγουμε αλληλευτικά προϊόντα. Ε, η, οι αλληλευτικέ μα δραστηριότητε συνδέονται άμεσα με τι άλλε δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. οι ψαράδε, οι αλληλεί συμβιώνουν με άλλες ε, χρήσεις, ε, λιμάνια, στρατιωτικές χρήσεις κλπ. που τους ε, περιορίζουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές. Οι εξορίξεις άμμου και άλλων στοιχείων από τη θάλασσα έγιναν στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών διαβούλευσης που όμως η, α, όπου όμως οι αλείς δεν ακουγόντουσαν τόσο πολύ όσο θα ήθελαν. Σε ό,τι αφορά ε, την ψυχολογία και τον τουρισμό στις παράκτιες ε, ζώνες, ε, για την ε, Μετροπολιτική Γαλλία είναι σημαντική δραστηριότητα. Ε, πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ ε, αντιπροσωπεύει η Αλία, περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ αντιπροσωπεύει η Αλία, αλλά η ψυχολογία και ο τουρισμό στι ίδιε ζώνε, στις ίδιες περιοχέ, τέσσερι φορέ περισσότερο, πάνω από τέσσερα δι δηλαδή. Ε, η συμβίωση με την ψυχαγωγία αρχικά δεν είχε δημιουργήσει προβλήματα στην, στους αλείς, αλλά ε, δεδομένης της των λιμένων ε, ή δεδομένες της ε, δημιουργίας ε, καινούριων ζωνών ψυχαγωγίας δημιουργήθηκαν προβλήματα. Οι καινούριες υποδομές και η οικιστική πίεση στις πράκτιες ζώνες ε, δημιουργούν πιέσεις ε, στο περιβάλλον και στους αλείς. Ε, η αεραστεχνική αλία από την άλλη μεριά ήταν πάντοτε προβληματική. όχι μόνο διότι δημιουργούσε πιέσεις στα αλληλευτικά αποθέματα, αλλά και γιατί δημιουργούν το πρόβλημα ανταγωνισμού σε περίπτωση πώληση των προϊόντων. Θα πρέπει αυτά τα πράγματα να ληφθούν υπόψη στο χωροταξικό συνδυασμό. Αυτό βέβαια θα το κάνει κάθε χώρα χωριστά. Σε ό,τι αφορά την ηχθειοκαλλιέργεια και την ανάπτυξή της, η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή ηχθειών από ηχθειοκαλλιέργεια είναι καλή. Το δε, τη δεχόμαστε. Αλλά να πούμε ότι οι ανησυχίε μας αφορούν την απέτηση υγειονομικής ασφάλειας και βιωσιμότητας αυτών των εξελίξεων στο μέλλον. Θα πρέπει να διατηρείται η καλή περιβαλλοντική κατάσταση του θάλασσιου περιβάλλοντος και να ακολουθούνται καλές πρακτικές, βέλτιστες πρακτικές. Η βιώσιμη διαχείριση ε, των ε, αποθεμάτων ε, που χρειάζονται για την τροφή των χθιοκαλλιεργειών είναι πολύ σημαντική. Άλλες δραστηριότητες, ε, όπως για παράδειγμα οι ανανεώσιμες πηγές στη θάλασσα κλπ, είναι πιο προβληματικές. Ε, ε, έχουν δημιουργηθεί καινούργιες ζώνες, για παράδειγμα προστατευμένες περιοχές, Natura 2000 κλπ. Οι αλληλείς δεν διαφωνούν υπό την προπόθεση ότι τα καινούργια σχέδια θα αποφασίζονται με διαβούλευση. Γι' αυτό το λόγο η Εθνική Επιτροπή μας έχει για τέτοιου είδους δραστηριότητες που επηρεάζουν την ε, αλία ε, έχει εκδώσει ιδιαίτερες ε, κατευθυντές γραμμέ. Είναι στη διάθεσή σας. Ο στρατηγικός προγραμματισμός βρίσκει σύμφωνους τους αλληλείς διότι τους εξασφαλίζει συμμετοχή στην χρήση του χώρου τάση ε, είναι ε, ο πολλαπλασιασμός των ε, δραστηριοτήτων στη θάλασσα, κάτι που περιορίζει τους αλλοίς. Γι' αυτό το λόγο επιθυμούν να γίνει ο χωροταξικός σχεδιασμός. Θεωρούν απαραίτητο οι ειδικές τους αλληλευτικές ζώνες να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία με την δημιουργία ζωνών λιγότερων περιορισμών για την αλία ε, και για τους επαγγελματίες αλληλείς. Με την χρήση, για παράδειγμα, καινούριων εγκαταστάσεων, μάλλον όταν δημιουργούνται νέες εγκαταστάσεις, ε, θα πρέπει κάθε φορά να διαβουλευόμαστε για να βρούμε ποιες είναι οι περιοχές της ε, που θα μπορούν να αφιερωθούν στην αλία με πολύ λίγους περιορισμούς. Ο γεωγραφικός καθορισμός ζωνών είναι πολύ σημαντικός και για τους ελείς όπως και για την ηθιοκαλλιέργεια. Σε ό,τι αφορά την θέση μας για τις δραστηριότητες, τις εξορρυκτικές δραστηριότητες, ε, η διαπίστωση είναι η εξής, απλή. Ε, οι τέτοιου είδους εκμεταλλεύσεις ε, εξορισμού δεν είναι βιώσιμες σε ανθρώπινη διάσταση, διότι κάποια στιγμή τα αποθέματα εξαντλούνται, δεν αναγεννώνται. Συνεπώς χρειάζονται, χρειάζεται να ακολουθούν οι πιο φιλικές προς το περιβάλλον στρατηγικές σε διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επιλογή των ε, περιοχών εξόρυξης και των τεχνικών εξόρυξης. Ο στρατηγικός σχεδιασμός αυτών των εξορυκτικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να γίνει με ε, καθορισμό συγκεκριμένων ποσοτήτων που θα είναι απολύτως απαραίτητες ε, και όχι περισσότερο και, η και με την ανακύκλωση των υλικών που εξάγονται και δεν χρησιμοποιούνται, εξορίσονται και δεν χρησιμοποιούνται. Αυτές οι εκμεταλλεύσεις είναι πολιτικές επιλογές που τροποποιούν και επηρεάζουν άμεσα το περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά σαν ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας στη θάλασσα, ε, μία απέτηση για τη χρήση τους είναι και πάλι η διαβούλευση με του αλληλεί, προκειμένου να επιλεγούν ή περιοχές που θα έχουν τη μικρότερη δυνατή επιπτώση στην Αλία. Έχουμε ήδη τέτοιου είδους διαβουλεύσεις στην Γαλλία με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το ίδιο και για την εγκατάσταση οποιασδήποτε ανεμογέννητρες κλπ. Σε ό,τι αφορά την, ε, τον καθισμό προστατευόμενων ζωνών, η υπερβολοντική ε, πολιτική ε, ε, επιβάλλει, όπως και η οδηγία πλαίσιο της Κομισιόν, ναι, καθορισμό νέων ζωνών ε, και την οργάνωσή του, την κατάλληλη οργάνωσή του Οι οργανώσεις των αλλιών θα πρέπει να θεωρηθούν ως βασικός φορέας επιτυχίας αυτής της διαδικασίας. Χρειάζεται ένα αποτελεσματικό εργαλείο που θα επιτρέπει την ε, την επιτυχία της εφαρμογής της 56-2008. Ε, ε, Έτσι ώστε και οι αλληλείς και οι θεοκαλλιεργητές ε, να έχουν τη δυνατότητα να χαίρουν του περιβάλλοντος στην κατάλληλη, στην, οικολογικά στην κατάλληλη κατάσταση. Έχουμε τέτοια παραδείγματα στη Γαλλία. Ε, έχουμε δει μικρές φώκες στην ε, Γαλλία οι οποίες είχαν δηλητηριαστεί ε, από φυτοφάρμακα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύ επηρεάζονται, επηρεάζεται το θαλάσσιο περιβάλλον. Τέλος, η σχέση με το δικαίωμα χρήσης. Η εγγύηση του συλλογικού δικαιώματος χρήσης είναι η βάση για μια κοινή διαχείριση κοινών πόρων. Έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα. Ε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ε, την απουσία ε, νομικής κατοχήρωσης των δικαιωμάτων των αλλιών να συνεχίσουν τις δραστηριότητε τους εκεί που παραδοσιακά τις τις ασκούν. Αυτό είναι μια δυσάρεστη διαπίστωση. Ε, σε άλλες ε, χώρες έχουν, έχει γίνει αναγνώριση των δικαιωμάτων των ε, ντόπιων ε, πληθυσμών. Ε, βρισκόμαστε πριν στην ίδια κατάσταση. Θεωρούμε ότι ενδεχομένως χρειάζεται να αναγνωριστούν τα παραδοσιακά δικαιώματα των αλλιέων. Αυτή η αναγνώριση των δικαιωμάτων στην εκμετάλλευση συγκεκριμένων περιοχών μπορεί να γίνει μέσω των ε, περιφερειακών ε, συμβουλευτικών επιτροπών. Η επιλογή, συγγνώμη, μέσω των ε, περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων, των ΡΑΚ. Τα ΡΑΚ έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο συσπήρωσης και διαχείριση του τομέα. Να σας πω τέλος, να σας υπενθυμίσω ότι η Διεθνής Ένωση Διατήρησης της Φύσης ε, είχε επιστήσει την ε, προσοχή μας στην Αυστραλία το 2005 στο γεγονός ότι ε, θα πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε ε, οποιαδήποτε περιβαλλοντική ή κοινωνικο-οικονομική ε, δράση η οποία θα διενεργείται χωρίς σεβασμό στους υπόλοιπους και θεωρώντας ότι τα ξέρουμε όλα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεντέλ. Με μεγάλο ενδιαφέρον πρόσεξα ότι σε όλες τις παρουσιάσεις το πρώτο τμήμα, κυρίως ε, στην παρουσίαση της κυρίας Μοντέζη και τώρα του κυρίου Κεντέλ, Αυτό που μας ενδιαφέρει ήταν να συμμετέχουν οι ενδιαφερέμενοι στο θαλάσσιο χωροταξικό ε, σχεδιασμό και να διαβουλευτούμε και με τους ίδιους τους ΕΛΕΗΣ. Δυστυχώς από την προσωπική μου πείρα στην Σκοτία δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και πολύ συχνά υπάρχουν προτάσεις για προστατευόμενες περιοχές ε, και απλώς κάποιος ε, τραβάει γραμμές σε ένα χάρτη και λένε στους αλληλείς ότι αυτή θα γίνει προστατευμένη περιοχή, πέρα τεράστιες περιοχές στη θάλασσα, χαράσσονται σε ένα χάρτη απλώς και μόνο για τους ε, σκοπούς της παράκτειας αιωλικής ενέργειας. Υπάρχει μια συγκεκριμένη περιοχή στη Σκωτία όπου υπάρχει μια πρόταση για τη δημιουργία του μεγαλύτερου αιωλικού πάρκου ε, παγκοσμίως, παράκτιο αιωλικό πάρκο ε, και υπήρχε ένα κείμενο 70.000 ε, σελίδων, ε, ζήγησε ένα τόνο και εγώ υπολόγισα ότι σε ένα δημόσιο υπάλληλο θα χρειαστεί 3,5 χρόνια να ε, διαβάσει αυτή την αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να εκπλήξει κανέναν το γεγονός ότι μπορεί να προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα και μετά από 10 χρόνια θα έρθει κάποιο και θα μας πει ότι εξαφανίστηκαν τα δελφίνια και οι υπόλοιποι ε, πανίδα της περιοχής και θα πει κάποιος από τις οικολογικές οργανώσεις μας να το είχαμε πει αυτό στη σελίδα 69.702 ε, που κανένας φυσικά δεν θα έχει καταφέρει να τη διαβάσει. Και νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι ε, αρνούμαστε ουσιαστικά την όλη δημοκρατική διαδικασία. Αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται μια συζήτηση για μια οδηγία για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και τα θέματα αυτά. Ε, το όλο θέμα όμως της διαβούλευσης από κάτω προς τα πάνω, διαβούλευσης με τον κλάδο, είναι κάτι το οποίο κατά την άποψή μου θα πρέπει να εξετάσουμε... και θεωρώ ότι η οδηγία αυτή μας δίνει την ευκαιρία να το κάνουμε. Ε, γνωρίζω και μια άλλη περίπτωση στις ακτές της Αγγλίας, στο Humberside, όπου υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα ανάπτυξης αιωλικής ενέργειας ε, που απειλεί ίσως τον καλύτερο αστακό σε όλη την Ευρώπη. Ε, μια περιοχή που παραδοσιακά παράγει αστακούς και καβούρια και έχει θρέψει ε, και βοηθήσει γενιές ολόκληρες αλλιέων. Και η κατασκευή αυτού του αιωλικού πάρκου θα μετακινήσει τόσες χιλιάδες τόνους άμμου που θα αλλάξει τελείως ε, ο βυθός της θάλασσας ε, στον οποίο θρέφονται οι αστακοί και τα καβούρια και, και στη συγκεκριμένη περίπτωση κανένας δεν μίλησε με αυτούς που αλλιεύουν αστακούς και καβούρια. Απλώς αποφασίστηκε ότι θα προχωρήσει το πρόγραμμα. Αυτό που μου κίνησε την περιέργεια είναι ε, το γεγονός ότι η κυρία Μοντέζη είπε ότι για ένα αλληλικό πάρκο μπορεί να χρειαστούν 8 μήνες για να δοθεί απλώς η άδεια, ενώ για μία ηχθειοκαλλιέργεια μπορεί να πάρει και δύο χρόνια η άδεια. Και είπατε κι εσείς ότι έστω και ένα μικρό ποσοστό αλευμάτων που θα μπορούσαμε να δώσουμε αντί να χρειαστεί να τα εισάγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιουργήσει πάμπολες θέσεις εργασίας. Ενώ στα αεολικά πάρκα υπάρχουν κάποιες λίγες θέσεις στη διάρκεια της κατασκευής, ένα-δυο άτομα για τη συντήρηση και αυτό είναι όλο. έχει δημιουργηθεί ολόκληρος δόρος για αυτά τα παράκτια ολικά πάρκα. Κατά την άποψή μου πρόκειται για μια ψευδοοικονομία η οποία είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και δεν θα είχε ποτέ επιβιώσει χωρίς τις επιδοτήσεις. Ε, και νομίζω ότι αυτό ε, ε, εκτοπίζει τους αλληλείς από παραδοσιακούς χώρους τους οποίους αλλιεύουν. Και ε, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν παγκοσμίω εκτοπίζουν επίση αλληλεί. Και τώρα που άκουσα και τον κύριο Κεντέλ, ο οποίο αναφέρθηκε στι ε, τεράστιε οικονομικέ πιέσει ε, για την θάλασσα και το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θεωρώ ότι αυτά απειλεί και τις μελλοντικέ γενναίες αλλιέων, αλλά και τις σημερινές γενιές. χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν για τις παρουσιάσεις αυτές. Καλημέρα σας κύριε Πατραονέβες. Ετοιμαζόμουν να πω ότι ανησυχώ λίγο που δεν είναι εδώ οι ομιλητές για το επόμενο τμήμα του πάνελ, αλλά με χαρά διαπιστώνω ότι η Μαρία Πατραονέβες είναι εδώ. Ε, είχαμε και αυτή την ε, ολονύκτια διαπραγμάτευση για τη μεταρρύθμιση της κοινή ελευθερικής πολιτικής. Ε, θέλει κανείς άλλος να σχολιάσει πριν ε, προχωρήσουμε στο επόμενο πάνελ. Οι ομιλητές και κυρία Τομάς, μήπως θέλετε να σχολιάσετε αυτά τα οποία είπα ή σας αρκούν. Κύριε Τομάς. Ναι, να ευχαριστήσω καταρχάς τους δύο μιλητές και όπως και εσείς κύριε Πρόεδρε με εξέπληξαν όλες αυτές οι προτάσεις και θα χρησιμοποιήσω και τη φράση του κυρίου Κεντέλ ε, αν γίνονται πράγματα χωρίς κανένα σχεδιασμό, χωρίς καμία διαβούλευση και χωρίς κατάλληλη διαχείριση των παράκτιων περιοχών, ελοχεύει ο κίνδυνος ε, να βρεθούμε σε μια κατάσταση ζούγκλας, ε, την οποία παρουσιάσετε κι εσείς ε, πολύ καλά ε, με αυτά τα οποία συμβαίνουν στις ακτές της Σκοτίας. Ε, και εμείς στη Βρετάνη έχουμε μια αντίστοιχη κατάσταση. Δηλαδή, αυτοί που ασχολούνται με την ενέργεια έχουν ε, ξεκινήσει η κατασκευή του πρώτου παράκτιου αιωλικού πάρκου στην πιο σημαντική περιοχή όπου έχουμε χτένια και ε, πραγματικά αυτά δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη κατά το σχεδιασμό τους και δεν λαμβάνονται μέτρα για να αποφευχθούν αντίστοιχες ε, καταστάσεις. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός θα είναι ένας τρόπος για να ρυθμίσουμε τη χρήση των χώρων και θα πρέπει να γίνει φυσικά και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το πρώτο τμήμα. Να περάσουμε τώρα στο δεύτερο πάνελ. Ε, ευκαιρίες για την αλία και την υδατοκαλλιέργεια και ε, δίνω με τα χαράς ε, το λόγο στην αγαπητή συνάδελφο την κυρία Μαρία Πατραονέβες για την εισαγωγή σε αυτό το τμήμα. after a horrible minute you were leaving. So. Κάποια στιγμή φοβήθηκα ότι φεύγεις. No, Mr. President, I'm not leaving. Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν φεύγω, μόλις έφτασα. Να ξεκινήσω ζητώντας συγγνώμη. Ήμουνα σε άλλη επιτροπή. Έτσι είναι η ζωή εδώ. Τρέχουμε από τη μία επιτροπή στην άλλη. Και απλά ήθελα να μιλήσω με τον επόμενο μιλητή, ώστε να βεβαιωθώ ότι όλα είναι έτοιμα για τις επόμενες παρουσιάσεις. Καταρχήν να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά να συμμετέχω σε αυτή την σημαντική ακρόαση που έχει να κάνει με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και που πρόκειται για μια ευκαιρία στην, ε, στις, ε, στην Αλία και στην Ιθιοκαλλιέργεια. Ο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό έγινε προτεραιότητα λόγω των πολλών διαφορετικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σήμερα στι θάλασσε και στου ωκεανού. Όπω όλοι ξέρουμε, από την αρχή τη ανθρωπότητα η θάλασσα πάντα ήταν πηγή τροφής και τρόπος μεταφοράς. Σήμερα όμως είναι επίσης ε, το τόπος ηχθειοκαλλιέργειας, δημιουργίας αιωλικών πάρκων, ε, κατασκευών, ε, τουρισμού και πολλών άλλων δραστηριοτήτων, ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Με τόσο πολλές διαφορετικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη θάλασσα, που συχνά ανταγωνίζονται για τον ίδιο χώρο ή παρεμβαίνουν η μία στην άλλη, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός πράγματι έχει γίνει προτεραιότητα. Πρόκειται για την ανάγκη να οργανώνονται όλες οι θαλάσσιες ε, δραστηριότητες ανάλογα με τις ανάγκες τους και ε, ανάλογα με τις ε, πιθανές επιπτώσεις της μιας δραστηριότητας πάνω στην άλλη. Στόχος είναι λοιπόν να επιτρέψουμε σε κάθε μια από αυτήν την ε, δραστηριότητα να αναπτύσσεται χωρίς να επηρεάζει αρνητικά τις άλλες και να αποφύγουμε ε, οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση. Ταυτόχρονα, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ε, προωθεί καλύτερη χρήση των πόρων ανθρώπινων, τεχνικών, οικονομικών και συμβάλλει με αποφασιστικό τρόπο στη βιωσιμότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Όσον αφορά την αλληλεία και την ηχθειοκαλλιέργεια, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός μπορεί να συμβάλλει στον ρόλο κλειδί που παίζουν οι δραστηριότητες αυτές. Ε, στις ε, θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, δημιουργώντας ε, νέες περιοχές για ηχθειοκαλλιέργεια ανάλογα με τα σχέδια που θα ετοιμαστούν από τα κράτη-μέλη, χωρίς να επηρεάζονται οι παραδοσιακές δραστηριότητες αλληλείας και μάλλον μοιράζοντας ε, τους ε, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι. Επίσης, ε, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός συμβάλλει σε οικοσυστημική προσέγγιση που θα συμβάλλει σε καλή ανάπτυξη και βιωσιμότητα της αλίας και της ηχθειοκαλλιέργειας. να πω με λίγα λόγια ότι ε, η ολοκληρωμένη εικόνα, η κατανόηση της ε, αλληλεπίδρασης και η ε, προώθηση των δυνατότητων συνέργειας είναι κάτι που θα συμβάλλει στην παρούσα και μελλοντική βιωσιμότητα των θαλασσών. Και στην ακρόαση αυτή έχουμε διάφορα πάνελ ε, που θα μας παρουσιάσουν διάφορες προσεγγίσεις ε, στο ίδιο θέμα. Εμείς θα επικεντρωθούμε στις ευκαιρίες ε, για την αλληλεία και την καλλιέργεια. Θα δώσω τον λόγο στον καθηγητή Ρικάρδο Σεράου Σάντος, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στις Αζόρες, καθώς και πρόεδρος της ΕΜΑΡ και θα μας μιλήσει για... Συγγνώμη. Κάποιος μου έδωσε έναν τίτλο τον οποίο δεν μπορώ να διαβάσω. Διαχείριση της, ε, της αλληλείας ε, και των ομάδων ε, στις, στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Έχει γίνει μια προσαρμογή στον τίτλο σε σχέση με αυτό που έχετε εσείς στο δικό σας πρόγραμμα. Ρικάρδο, έχεις το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή και τη δυνατότητα να συζητήσω εδώ θέματα ε, θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Θα επικεντρωθώ στις Αζόρες. Και θα ε, αναφέρω ότι η ηχθειοκαλλιέργεια ακόμα δεν είναι θέμα στις Αζόρες. Οι Αζόρες είναι το όπως όπου η εμπορική και αλληλεία και η ε, αλληλεία αναψυχής ε, είναι πολύ μεγάλη σημασία. Είναι ε, μια ιδιαίτερη γεωγραφική περιοχή. Και επίσης ε, επίκειται στο εγγύς μέλλον υποβρύχια εξόριξη με μετάλλων. Το 94% του βυθού είναι πάνω, έχει βάθος ε, μεγαλύτερο των χιλίων μέτρων και ε, υπάρχουν εδώ ευάλωτα οικοσυστήματα. Ε, έχουμε κοράλια ψυχρών υδάτων και έχουμε κάποια είδη προτεραιότητας όπως είναι κάποιοι καρχαρίες του βυθού και διάφορα άλλα φαλαινοειδή. Ε, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι ένας από τους τρεις πυλώνες ε, της Εθνικής Στρατηγικής Θαλάσσης που έχει υιοθετηθεί από το 2004. Υπάρχει μια μακρά ε, παράδοση προστασίας διαφόρων ειδών στις αζόρες και των οικοσυστημάτων τους όπως είναι οι καρχαρίες. Ε, αυτά τα σχέδια αποτελούν σημαντικό στοιχείο της, ε, του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και των ε, πολιτικών διατήρησης. Η διαφάνεια που βλέπετε τώρα θα μπορούσε να είναι η τελική μου δήλωση, αλλά οι μελέτες που έχουμε κάνει στις Αζόρες καταλήγουν ότι το κοινό στις Αζόρες και έχουν γίνει διάφορες μελέτες σε, σε διάφορους τομείς της κοινωνίας. Το κοινό αντιλαμβάνεται ε, την, ε, τους στόχους διατήρησης ε, με την ευρύτερη έννοια. Δηλαδή κοιτάει πέρα από το ένα είδος και διαπιστώνει ότι υπάρχει σημαντικό όφελος με τη διατήρηση των ειδών και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για την διατήρηση μιας σειράς ειδών παρά για την διατήρηση ενός είδους μόνο. Του ενδιαφέρει δηλαδή ε, το σύνολο του οικοσυστήματος ε, και αυτό προέρχεται από μια παράδοση ε, ουσιαστικά θαλάσσιο χωροταξικού σχεδιασμού στις Αζόρες. Σε Αζόρες λοιπόν έχουμε νησιά και υφάλους και η ύφαλοι αυτή ε, ε, είναι πολύ σημαντική ε, για το οικοσύστημα. Ξέρουμε ότι πολλά από τα πελαγικά είδη καρχαρία συχνά συγκεντρώνονται εκεί. Και μεγάλο μέρος της αλίας αφορά τον... τον έχουμε τις θαλάσσιες χελώνες. Αν κοιτάξουμε την ε, την κίνηση των ε, θαλάσσιων ε, χελώνων βλέπουμε ότι ο αριθμός των ημερών που περνούν κοντά στους υφάλους είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των ημερών που περνούν στα ανοιχτά του ωκεανού. Και έχουμε πολύ καλή περιγραφή τώρα πια των, οικοσυστημάτων, ε, των θαλάσσιων οικοσυστημάτων ε, στις Αζόρες. Ε, σας είπα ότι έχουμε περίπου 500 υφάλους, έχουμε κοράλια και μάλιστα με περισσότερα από 166 διαφορετικά είδη Έχουμε διάφορους, ε, διάφορα είδη οικοσυστημάτων ε, που ε, αποτελούν προτεραιότητα και σε ευρωπαϊκές και σε διεθνείς συμβάσεις. Η αλία στις Αζόρες έχει παρουσιαστεί σε έγγραφο των συναδέλφων μου Χριστοφάν και Τερμομοράτο. Και Η μελέτη αυτή δείχνει ότι τη δεκαετία του 50 η αλληλεία αφορούσε κυρίως ε, τα ε, ε, μεγάλα κοιτοειδή. Αλλά λόγω της νομοθεσίας και λόγω της μείωσης του τομέα αυτού, βλέπουμε ότι η αλληλεία κυρίως επηρεάζεται από τη διακύμανση των πελαγικών ειδών και διαπίστωσαν ότι η αλληλεία στις αζόρες έχει αυξηθεί όσον αφορά τα διάφορα είδη στόχη. Και με την καλύτερη συνεννόηση μεταξύ επιστημόνων, αλλιέων και των αρχών, με την καλύτερη διαχείριση της αλληλείας, προσεγγίζουμε τώρα τον σωστό αριθμό αλλιευμάτων, διότι στο παρελθόν πολλά από τα είδη αυτά ε, δεν καταχωρούνταν διότι μιλούσαμε για ένα είδος ενώ στην ουσία πρόκειτο για διαφορετικά είδη. Κάτι άλλο όμως που διαπιστώνουμε και που δείχνει αυτή η μελέτη είναι ότι μειώνεται ο αριθμός των ε, ψαριών που ε, παίρνουμε από τη θάλασσα λόγω των ποσοστώσεων και των τάκ. Όλα αυτά επηρεάζουν σημαντικά την αλληλεία. Και επίσης βλέπουμε τον χώρο εδώ πέρα που καταλαμβάνει ο στόλος. Σε πράσινο πρόκειται για τον εθνικό και περιφερειακό στόλο. Με κόκκινο βλέπετε ε, τα άλλα ευρωπαϊκά σκάφη, αλλά ουσιαστικά βλέπουμε όλοι, όλος ο χώρος καταλαμβάνεται αυτή τη στιγμή. Εδώ βλέπετε την ε, πελαγική και βενθοπελαγική αλληλεία. Ε, σημαντικό στην ε, αλία στην περιοχή είναι η αλία βυθού ε, σε βάθος 500 έως 1500 μέτρων. Και ενώ έχουμε μία τεράστια αποκλειστική οικονομική ζώνη έκτασης ενός εκατομμυρίου τετραγωνικών χιλιόμετρων, μόνο μέρος της είναι κατάλληλο για αλληλεία. Και βλέπετε ότι η περιοχή αυτή όπου γίνεται η αλία αυτού του τύπου είναι ακριβώς ε, η, η, η περιοχή με τα ευάλωτα οικοσυστήματα όπως είναι τα κοράλια. Βλέπετε λοιπόν εδώ τις ε, διάφορες ε, ε, ταξονομικές ομάδες κοραλιών Υπάρχει λοιπόν ε, μεγάλη σχέση ανάμεσα στα, ε, στα ψάρια και στα ευάλωτα οικοσυστήματα. Γιατί είναι ευάλωτα τα οικοσυστήματα αυτά. Ε, πρέπει να κοιτάξουμε την ηλικία των οργανισμών αυτών. Ε, κάποιοι οργανισμοί φτάνουν σε ηλικία 3.000 ετών. το ζώο αυτό βλέπετε είναι αντικείμενο μιας μελέτης που που παρουσιάστηκε ε, το 2013 γεννήθηκε το 1192. Ε, έχουμε ε, λοιπόν, κάποια κοράλια, κάποια οικοσυστήματα τα οποία επιδοτούνται με το πρόγραμμα πλαίσιο 7 ε, βλέπουμε ότι η βιομάζα των ψαριών ε, ε, συνδέεται ε, είναι ανάλογη, είναι απευθείας ανάλογη με τα κοράλια και τα οικοσυστήματα αυτά. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε αυτή τη διαφάνεια. Η μελέτη αυτή <clears throat> στόχο έχει να σας δώσει μια επισκόπηση ε, των ε, οικολογικά και βιολογικά σημαντικών υφάλων ε, στην περιοχή. Βλέπουμε ότι Βλέπουμε ότι οι περιοχές που είναι πιο πιθανό να ονομαστούν βιολογικά και οικολογικά σημαντικές ε, απειλούνται σημαντικά. Ένας από τους ε, καλούς υφάλους ε, προστατεύεται με τη Συμφωνία των Αλλιέων στις Αζόρες. και είναι μια περιοχή όπου υπάρχουν πολλά καθρεφτόψαρα. Οι δραστηριότητες που ξεκινούν τώρα αφορούν τα πολυμεταλλικά θιούχα και ε, υπάρχει λοιπόν ε, αυτή η προσπάθεια, δεν τα βλέπετε αυτά ε, εδώ στην στην διαφάνεια, αλλά υπάρχει χαλκός, υπάρχει ψευδάργυρος, χρυσάφι. Κυρίως μας ενδιαφέρει ο χαλκός εδώ. Και πρόκειται για μια περιοχή για την οποία έχει συναυθεί σύμβαση με την εταιρεία ε, Ναυτίλος. Και έχουμε τρεις προστατευμένες περιοχές ε, για ε, επιστημονικούς ε, στόχους ε, και το πρόγραμμα Ναυτίλος μας ζητάει ακριβώς τις περιοχές αυτές. Άλλο θέμα που μας ενδιαφέρει στη διαχείριση της θάλασσας και του βυθού είναι οι διάφορες ρυθμιστικές αρχές. Βλέπετε εδώ την περιοχή ICS, βλέπετε την αποκλειστική οικονομική ζώνη, καθώς και κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2005, που απαγορεύει ε, οτιδήποτε που να ε, βλάπτει τα ε, οικολογικά οικοσυστήματα, τα ευάλωτα οικοσυστήματα εδώ πέρα, όπως είναι οι τράτες βυθού, οι σειρώμενες τράτες βυθού. Το 2011 έχουμε το θαλάσσιο πάρκο των Αζόρων, που καλύπτει έκταση, δεν έχω εδώ δεν έχω εδώ ε, το, το, τον ακριβή αριθμό, αλλά καλύπτει πάνω από 100.000 ε, ε, τετραγωνικά χιλιόμετρα που περιλαμβάνει προστατευόμενα νησιά, δύο, σημαντικά οικοσυστήματα, δύο περιοχές σημαντικές για τα πουλιά, για τα πτηνά, αυτό όμως ε, είναι το 1% της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και το 0,5% ε, του βυθού. Αποτελεί όμως ε, μεγάλο ποσοστό του βυθού με βάθο άνω των χιλίων μέτρων. Τα μέλη της ΟΣΠΑΡ υιοθέτηση είναι απόφαση για προστασία της ε, στήλης ύδατος ε, στην ε, περιοχή αυτή του μέσω Ατλαντικού βόρεια των Αζόρων. Και η προστασία των ευαίσθητων αυτών οικοσυστημάτων δείχνει ότι το 15,3% περιλαμβάνουν πάνω από 15 είδη και ομάδες ε, κοραλιών ε, βαθέων υδάτων. Πιστεύω λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο ε, όσον αφορά την προστασία των διαφορών ποικιλιών των κοραλιών. Η κατανόηση των κοινών ε, αξιών όσον αφορά την ε, βιοπικιλότητα και την ε, προστασία της θάλασσας. Ήταν αντικείμενο μελέτης που έγινε στην Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Αζόρες και δείχνει ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για τη βιοπικιλότητα. και βλέπουμε εδώ ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός ε, σχεδιασμός ε, αποτελεί σημαντικό εργαλείο. Η άλλη αυτή μελέτη που βλέπετε στην οθόνη που ε, δημοσιεύτηκε νομίζω φέτος ή στο τέλος της περσινής χρονιάς. Δηλαδή, η διαχείριση που βασίζεται στα οικοσυστήματα θα πρέπει να προωθηθεί ως ε, επιτυχημένη δημόσια πολιτική. Χρειάζεται όμως ε, συμμετοχή των πολιτών. Ε, θα πρέπει να δημιουργηθεί κοινωνικό κεφάλαιο ώστε να υπάρχει πιο αποτελεσματική και δίκαιη διαχείριση των θαλασσών της Ευρώπης. Το συγκεκριμένο αυτό συμπέρασμα συνδέεται με μία διαφάνεια του πρώτου ομιλητή, ε, της πρώτης ομιλητής εδώ σήμερα. Είπε ότι ακόμα εισάγουμε το 65% ε, των ε, ψαριών και θαλασσινών. Και από πού προέρχονται όλα αυτά. Από τόπους όπου δεν υπάρχει καλή ρύθμιση για την αλληλεία ούτε για την χθιοκαλλιέργεια. Και γι' αυτό ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ακόμα ποιες είναι οι επιλογές τους ε, όσον αφορά την προστασία της βιοπικιλότητας ε, και, ποια θα, και τι είναι προς όφελός τους, διότι εισάγουμε ψάρια τα οποία ε, προέρχονται από προβληματικά αλιευτικά αποθέματα. Και αυτό είναι κάτι που σκέφτηκα όταν, όταν είδα την ε, διαφάνεια. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ε, Ευχαριστούμε, Ρικάρδο. Θα δώσω το λόγο αμέσω στον επόμενο μιλητή. Και μετά θα σας καλέσω εδώ για να ε, ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θα ακούσουμε τον Πιέρ ε, Κάρλισκίντ. Είναι εδώ. Α, ωραία. Θα μείνετε εκεί στη θέση σας ή θέλετε να έρθετε εδώ. Εκεί, ωραία. Δεν είμαι σίγουρος, σίγουρη ότι διαβάζω σωστά το όνομά σας. Ε, Κάρλισκίντ θα μας, θα μας πείτε εσείς πώς είναι το όνομά σας, πώς διαβάζετε. Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Βρετάνης. Θα μας μιλήσει για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών, ε, ευκαιρίες για την αλία και την ηχθειοκαλλιέργεια. Ο πρώην ομιλητής μίλησε μόνο για την αλία, τώρα θα ακούσουμε μερικά πράγματα και για την ηχθειοκαλλιέργεια και μετά θα ακολουθεί συζήτηση ελπίζω ενδιαφέρουσα και για τις σχέσεις ανάμεσα στον αλληλευτικό τομέα και την ηχθειοκαλλιέργεια. Έχεις το λόγο. Merci. Ε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ας υπογραμμίσουμε καταρχήν ότι με χαρά βλέπουμε που η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται πολιτικές υπέρ της ε, θάλασσας και των παράκτητων περιοχών. Ε, το έγγραφο εργασίας ε, δείχνει ότι η θάλασσα αποτελεί σημείο εστίασης των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές, διαφορετικά έθιμα ε, στα κράτη-μέλη και είναι σημαντικό όλα αυτά να τα συνδυάσουμε ε, για να διασφαλίσουμε όλες τις δραστηριότητε στη θάλασσα και όλους τους φορείς αυτών των δραστηριοτήτων. Είναι πολύ δύσκολο η Ελία να αποκοπεί από το πλαίσιο μιας συνολικής ε, διαχείρισης των θαλάσσιων περιοχών, των παράκτιων περιοχών η ολοκληρωμένη διαχείριση θα πρέπει να θεωρείται ως ε, ορισμός και η εφαρμογή μιας ε, πολιτικής ε, βιώσιμης ανάπτυξης σε ένα συγκεκριμένο μέσο που είναι σε μια συγκεκριμένη περιοχή που είναι οι παράκτιες περιοχές. Περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες και όλα τα συμφέροντα αυτών των περιοχών με στόχο να τα κάνει σύμβατα, να τις κάνει συμβατές μεταξύ τους ενώ ταυτόχρονα θα διατηρεί θα συντηρεί την λειτουργικότητες ε, ε, των περιοχών αυτών. Οι περιοχές αυτές είναι περιοχές σύγκλησης και συμβίωσης δραστηριοτήτων θάλασσας και, θάλα, και ε, Παρ' όλα αυτά, ο περιορισμός των 12 μιλίων στη θάλασσα είναι ένας περιορισμός λειτουργικός. Από την άλλη μεριά είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνουμε ένα παρόμοιο καθορισμό στην στεριά, γιατί στη στεριά οι δραστηριότητε, οι λειτουργίε ε, πηγαίνουν πολύ πιο μακριά μερικέ φορέ. Για παράδειγμα, η Βρετάνη θα έπρεπε συνολικά, με βάση την, τα γεωγραφικά τη χαρακτηριστικά, να θεωρηθεί ω ε, παράκτια περιοχή. Ε, ο χωροταξικό σχεδιασμός αποτελεί ένα εργαλείο της ε, συνολικής διαχείρισης. Η αποτελεσματικότητα και η χρηστικότητα του σχεδιασμού ε, εξαρτάται από το πώς γίνεται ε, θα πρέπει να βοηθήσει στην ε, λήψη αποφάσεων για την πρόσβαση στα σωρευτικούς πόρους και στις αλευτικές περιοχές. Ο χωροταξικός διαδρομός στη θάλασσα θα πρέπει να αποτελεί λοιπόν εργαλείο εφαρμογής των, ενός ιδανικού για τις περιοχές αυτές. Θα πρέπει αφενός η χρήση της ε, θάλασσας από τον άνθρωπο να μην δημιουργεί προβλήματα στη των οικοσυστημάτων και δεύτερον να, διασφαλίζουμε την, να διασφαλίσει την καλή συμβίωση των δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή ενός εργαλείου σχεδιασμού αποτελεί έκφραση μιας ε, πολιτικής ε, βούλησης. Χρειάζεται μια διακυβέρνηση που θα είναι ικανή ε, να μετατρέψει τους στόχους σε πραγματικότητα. Χωρίς την στενή σχέση ανάμεσα στο εργαλείο και την διακυβέρνησή του, ο χωροταξικός σχεδιασμό δεν είναι δυνατόν να πετύχει τους στόχους του. Το παράδειγμα του ε, θαλάσσιου πάρκου της Αρουάς δείχνει αυτό το, τη, της ήρωας συγγνώμη, δείχνει αυτό το αποτέλεσμα. Τα, ε, το χωροταξικό σχεδιασμό δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες λεπτομερείς ε, ε, χρήσεις, περιλαμβάνει κάποιες προτεραιότητες, απλώς όμως με κάποια ασάφεια. Πρόκειται για μια, ένα καθορισμό ζωνών που δεν ονομάζεται έτσι, αλλά η κατάσταση αυτή είναι ασαφής και μπορεί να δημιουργήσει πολλές συγκρούσεις. Επικρατεί ένα φλού για τις δραστηριότητες. Η αλία δεν απαγορεύεται, παρόλα αυτά είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς ε, πώς ακριβώς τη μορφή θα, λάβει. Είναι πολύ δύσκολο και για τους τοπικούς φορείς. το Συμβούλιο Διαχείρισης του Πάρκου δεν έχει, ε, δεν έχει αρμοδιότητες απόφασης, μόνο εκτελεστικές αρμοδιότητες. Ε, ε, και πολύ ε, συχνά δημιουργούνται ε, προβλήματα διότι δέχεται πιέσεις από τους φορείς να αντιστρέψει αποφάσεις. Ε, η παράκτια ζώνη είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να αντέξει τον παραπλησιασμό των χρήσεων στο δίνεκες. Θα πρέπει να γίνονται επιλογές με συγκεκριμένες προτεραιότητες δραστηριοτήτων. Δύο είναι τα σημεία κλειδιά στην εφαρμογή ενός χωροταξικού σχεδιασμού. Πρώτον, να έχουμε επαρκή γνώση, επαρκή στοιχεία, το είπαμε αυτό ήδη, και δεύτερον, μεθοδολογικά κριτήρια για τον καθορισμό προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες. Δεν θα, δεν θα επανελθώ στο πρώτο από αυτά. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, τα μεθοδολογικά κριτήρια, αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται περιβαλλοντικά κριτήρια. Για παράδειγμα, η οδηγία πλαίσιο στρατηγική για το θαλασσιο περιβάλλον. Όμω αυτή δεν είναι αρκετή. Αυτά τα κριτήρια δεν είναι αρκετά. Γιατί ε, ο στόχος είναι η ε, βιώσιμη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, συνεπώς χρειάζεται και ένας βιώσιμος σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός είναι και πάλι ένα εργαλείο ε, στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης, οπότε θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οικολογικά αλλά και κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Ε, η αξιολόγηση, στην αξιολόγηση ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων λοιπόν των δραστηριοτήτων θα πρέπει να προστίθεται και η αξιολόγηση των οικονομικών και κοινωνικών ε, ε, επιπτώσεων των δραστηριοτήτων. Χρειάζεται λοιπόν να μιλήσουμε όχι μόνο για οικολογικό ίχνος αλλά και για κοινωνικο-οικονομικό ίχνος. Ως τώρα λέγαμε, μιλούσαμε μόνο για το, οικονομικό, για το οικολογικό ίχνος. Δεν αρκεί αυτό γιατί δεν λαμβάνει υπόψη ε, την αλεξάρτηση των ε, περιοχών στις οποίες αναπτύσσονται οι δραστηριότητες. Το παράδειγμα της ε, Βρετάνης και του κόλπου του Μορμπιόν το αποδεικνύει αυτό. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαχείρισης το ε, στο αμυκτό συνδικάτο του κόλπου του Μορμπιόν ε, ξεκίνησε μια εργασία για να βελτιστοποιήσει τις ε, ε πρακτικές που ακολουθούνται για την αλία και την ε, ηχθειοκαλλιέργεια προκειμένου να τις εξισορροπήσει. Τα αποτελέσματα ήταν η εφαρμογή ενός συστήματος γεωγραφικής ε, Προγραφικού προσδιορισμού των ε, καλλιεργιών κοχυλιών ε, και ταυτόχρονο καθορισμό ζωνοναλίας. Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των, δραστηριοτήτων, των ανθρώπινων δραστηριοτήτων μας οδηγούν στο να κάνουμε επιλογές με βάση τρία κριτήρια. Ε, ο, πρώτον ο βαθμός αποκλειστικότητας και συμβίωση των δραστηριοτήτων. Αντίθετα με τις χερσές δραστηριότητες ε, που απαιτούν αυστηρή χωροταξία ε, και είναι δύσκολη η ανακατανομή του χώρου, στο, στο θαλάσσιο περιβάλλον δεν χρειάζονται πολλές υποδομές στη θάλασσα ε, και δεν είναι απαραίτητο η χρήση να είναι αποκλειστική. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε ανεμογεννήτρες, αιωλικά πάρκα και ταυτόχρονα αλεία. Ε, ή ε, καλώδια στο βυθό της θάλασσας και αλία Θα πρέπει να δούμε πώς είναι δυνατόν να συμβιώσουν δραστηριότητες χωρίς ε, να προσβάλλονται τα, τα οικολογικά συστήματα, τα περιβαλλοντικά συστήματα. Η κυρία Τόμας μίλησε για το αιωλικό πάρκο του Σέμπριγιό. Αυτό δείχνει ότι στο πλαίσιο της πολιτικής ανάπτυξης των ανασύμων πηγών ενέργειας η Γαλλία ε, καθόρισε ζώνες για αιωλικά πάρκα και στην Βρετάνη ένα από αυτά είναι το Saint-Brieuc, ε, σε μία από τις ε, περιοχές που χρησιμοποιούνται πιο πολύ από την Αλία. Απριόρι, ε, αυτά, αυτές οι δύο δραστηριότητες είναι συγκρουσιακές. Δημιουργούνται προβλήματα για την δημιουργία τέτοιων αερολικών πάρκων στη Βρετάνη. Σε συνεργασία με τους αλείς όμως έγινε μια δουλειά για να γίνουν συμβατές αυτές οι δύο δραστηριότητες. ήταν σημαντικό να δούμε ποιες είναι ε, οι πρακτικές των αλλιέων και αυτό επέτρεψε να ε, αλλάξουμε τα όρια έτσι ώστε να μπορούν μέσα στο αιωλικό πάρκο να συνεχίσουν, να συνεχιστούν οι αλληλευτικές δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο έγιναν συμβατές οι δύο δραστηριότητες. Ε, δημιουργήσαμε τεχνητούς υφάλους ε, πάνω στους οποίους στήθηκαν οι, ε, οι γεννήτρες και ταυτόχρονα σε αυτούς γίνεται και, γίνονται και δραστηριότητες αλίας. Με αυτόν τον ε, τρόπο καταφέρουμε να συνδυάσουμε τις δύο δραστηριότητες. Ο μιλητής μιλάει εξαιρετικά γρήγορα, δεν είναι δυνατόν να τον παρακολουθήσουμε. θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και η βιωσιμότητα ο χωροταξικό σχεδιασμό θα πρέπει να τη λαμβάνει υπόψη, ε, λαμβάνοντα υπόψη ταυτόχρονα και τη δυνατότητα αυτών των δραστηριοτήτων, ε, την εξέλιξη του μάλλον στο μέλλον. Μια δραστηριότητα δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη σημερινή τη ικανότητα, αλλά ε, τη μελλοντική τη. Οι αλευτικέ δυνατότητε είναι πολύ σημαντικέ, για παράδειγμα. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, τις επιπτώσεις των εργαλείων που χρησιμοποιούνται, τις συνθήκες υγιεινής κλπ. Και υπάρχει περιθώριο για τη βελτίωση της βιωσιμότητάς της, της αλληλευτικής δραστηριότητας. Αυτό γίνεται και στην Βρετάνη. Τέλος, ε, οι κανονισμοί που διέπουν τις δραστηριότητες στη θάλασσα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις, τις εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν, ε, και, τις, και τα λευτικά, ε, τους πόρους. Ε, για παράδειγμα, στην Βρετάνια έχουμε πολύ εξορρεκτική βιομηχανία, ε, οπότε υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από αυτήν της χώρας και θα πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη. Η αλληλεία έχει ένα σημαντικό μια σημαντική συνεισφορά στην τοπική οικονομία και στην τοπική κοινωνία. Τώρα έχουμε καινούριε δραστηριότητε και ταυτόχρονα την ανάπτυξη καινούριων ζωνών προστασία. Αυτά συναγωνίζονται, ανταγωνίζονται μεταξύ τους εις βάρος παραδοσιακών δραστηριοτήτων ε, που δεν κατάφεραν να ακουστεί η φωνή τους όσο πολύ θα ήθελαν. Γιατί αυτές οι καινούριες τεχνολογία για παράδειγμα είναι πολύ πιο πολλά υποσχόμενες. Θα πρέπει να ακούσουμε τη φωνή των αλλιέων, τη φωνή αυτών των παραδοσιακών δραστηριοτήτων. Η Βρετάνη ε, αποκτήσε την χάρτα των ε, ε παράκτιων περιοχών που ε, έχει περιλαμβάνει δίκτυα σχεδίων ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτηων περιοχών. Χρειάζεται λοιπόν ο χωροταξικός σχεδιασμό να πηγαίνει χέρι-χέρι με την ολοκληρωμένη διαχείριση. Σας ανέφερα ποια είναι τα κριτήρια για την ολοκληρωμένη διαχείριση, για το χωροταξικό σχεδιασμό. Τώρα να σας πω ορισμένα πράγματα για την οδηγία πλαίσιο. Ε, από μεθοδολογικής πλευράς, ο ε, η χωροταξικός δεν πρέπει να είναι μόνο χωροταξικός. Ε, θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα, ο καρπός μια σημαντικής δουλειάς ε, για τους πόρους και τις δραστηριότητες στη θάλασσα και έχουμε δύο συμπεράσματα για αυτό το θέμα. Πρώτον, ε, σε ό,τι αφορά την επιλογή μιας οδηγίας πλαίσιο. Δίνει εγγυήσεις, αλλά αφήνει στα κράτη-μέλη ε, τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τη δική τους μεθοδολογία. Το καταλαβαίνω αυτό. Τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές παραδόσεις, διαφορετικά έθιμα, Παρ' όλα αυτά αυτή η επιλογή αποτελεί και αδυναμία. Γιατί έχουμε δει παλιότερα ότι η επιλογή ενό χωροταξικού σχεδιασμού στη θάλασσα εξαρτάται πολύ σε μεγάλο βαθμό από τη μεθοδολογία. Δεύτερον, δεύτερη παρατήρηση συμπέρασμα, ε, η σύνδεση του χωροταξικού σχεδιασμού στη θάλασσα με την ολοκληρωμένη διαχείριση. Η ολοκληρωμένη διαχείριση είναι μια πολιτική αποφασιστικότητα με πολιτική βούληση. Συνεπώ, λαμβάνει υπόψη συμφέροντα, έχει στρατηγικού άξονε δράσει, και ένα σύστημα διακυβέρνησης. Ο χρεοταξικός σχεδιασμός στη θάλασσα την άλλη μεριά είναι ένα εργαλείο εφαρμογής και παρακολούθησης αποφάσεων που λαμβάνονται για την διαχείριση. Ε, συνεπώς έχουμε στο ίδιο επίπεδο ένα εργαλείο και μια ε, πολιτική βούληση. Θα πρέπει να καθοριστεί η διασύνδεση μεταξύ τους και η τους, η αλληλεπίδρασή τους. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Καρλέσκινς. Έβαλα και το σωστό τόνο, Καρλέσκινς. Μάλλον το είπα λίγο καλύτερα το όνομά σας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και οι δύο παρουσιάσεις. Μας δώσατε δύο παραδείγματα, ένα των Αζωρών ε, στον Ατλαντικό ωκεανό και το άλλο της Βρετάνης, ε, μιας παράκτιας περιοχής. Ο ένας ε, στάθηκε κυρίως στην ανάγκη μιας μεγαλύτερης εμβάθυνσης και ο άλλος αναφέρθηκε κυρίως στα μεθοδολογικά κριτήρια Με αυτό το διτό όραμα, καταφέραμε να δούμε ποιοι είναι οι δύο μεγάλοι τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούμε εάν θέλουμε να κάνουμε κατάλληλο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο τους ε, συναδέλφους, αλλά πριν ε, σας δώσω το λόγο θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής στους ομιλητές. Ξέρουμε ότι ο τίτλος ε, για το πάνω μας ήταν «Δυνατότητες για την αλία και την υδατοκαλλιέργεια». Δυνατότητες συνήθως σημαίνει κάτι θετικό και θα ήθελα να ξέρω από πλευρά σας, διότι ε, έχετε δύο ε, οπτικές οι οποίες συμπληρώνουν η μία την άλλη. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει για την αλληλεία σε αυτό το νέο εντό εισαγωγικών πρόγραμμα, αυτό το νέο πρόγραμμα του θαλάσσιου χωροτεξικού σχεδιασμού. Εμείς ε, ασχολούμαστε με τον τομέα της αλληλείας και θέλουμε πάντα να γνωρίζουμε τι δυνατότητες υπάρχουν για την αλληλεία ε, ποια είναι τα θετικά στοιχεία για την αλληλεία, αλλά υπάρχουν και άλλοι που με τον ένα με τον άλλο τρόπο αναμένουν αυτό το ε, θέμα του το θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού ως ένα τρόπο για να περιορίσουν, αν όχι και να καταβοραθρώσουν ακόμα περισσότερο, την αλία. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να ακούσω από εσάς τους δύο είναι το εξής. Ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά στοιχεία αυτού του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού για την αλία. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη ερώτηση και για τους δυο σας. Και στη συνέχεια θα δω αν υπάρχει κάτι, ε, κάποιος άλλος ο οποίος ε, θέλει τον λόγο. Ε, I in language I should... Δεν ξέρω τώρα σε ποια γλώσσα θα πρέπει να απαντήσω. Να μιλήσω αγγλικά, πορτογαλικά, χωρίς μικρόφωνο, πρόεδρε. ah, η πολυγλωσία είναι αναπόσπαστο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να μιλήσετε πορτογαλικά. Ε, θα προτιμήσω να μιλήσω πορτογαλικά. Λοιπόν, νομίζω ότι η αλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένας προβληματικός ε, κλάδος. τις Αζόρες οι το γνωρίζουν και υποστηρίζουν ε, μοντέλα χροταξικού σχεδιασμού, υποστηρίζουν τις ε, προστατευμένες αλευτικές, ε, θαλάσσιες ζώνες, γνωρίζοντας εξ αρχής διότι υπάρχουν ευρωπαϊκές ε, μελέτες. Εγώ με την Βανέσα πριν από κάποια χρόνια αξιολογούσαμε τη, τα ωφέλη και για την αλία των προστατευόμενων θαλασσίων ζωνών και γνωρίζουν ότι ε, οι αλίες ότι ε, ε, ε, τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα 20 χρόνια δεν φαίνονται σαφώς τα ωφέληματα, αλλά μετά ναι. Οι αλίες θα πρέπει να... Οι αλίες τα γνωρίζουν αυτά και υποστηρίζουν τέτοιου είδου ε, χωροταξικούς σχεδιασμούς τη θάλασσα. Αρχικά ζητούσαν επιδοτήσεις, αλλά τώρα πια βλέπουμε ότι δεν επιμένουν σε τέτοιου είδους αιτήματα. Διότι γνωρίζουν πως αργότερα θα προκύψουν ωφέλη και για αυτούς. Τώρα, κάτι που έχει ε, δημιουργήσει προβλήματα στο σύστημα είναι η προοπτικές αξιοποίησης ε, βιώσιμων μορφών αλίας, οι οποίες ε, ε, πλήττονται από πολιτικές, ε, εμπορικές πολιτικές ανοιχτών αγορών που αυξάνουν τις εισαγωγές. Ήρθε να προσθεθεί και η κρίση, η οικονομική κρίση και οι αλείς βλέπουν ότι διαψεύδονται οι ελπίδες τους να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία το προϊόν τους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο που μας ε, επηρεάζει και εμάς. Αυτή τη στιγμή ε, θέλουμε να ακολουθήσουμε μια πολιτική, μια λογική που να εστιάζεται στο οικοσύστημα, κάτι που οδηγεί και δημιουργεί ελπίδε για την βελτίωση τη αξία του προϊόντος, αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Νομίζω ότι ο πρώτος άξονας είναι να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας, όπως το υπενθυμίσατε κι εσείς, ε, είναι μία από τις σημαντικές προϋποθέσεις για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και ένα και από τα βασικά στοιχεία. Και όταν ε, μιλάω για βελτίωση των γνώσεών μας, σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζουμε και το περιβάλλον, αλλά και τις συνέπειες, τις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες ε, της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως σας έλεγα. Θα πάρω το παράδειγμα του κόλπου του Μελπιγιόν, όπου έχουμε υδατοκαλλιέργεια. Έχουμε όμως υδατοκαλλιέργεια και εκθοκαλλιέργεια και στη Βρετάνη και σε άλλες περιοχές. Είναι παραδοσιακές δραστηριότητες αυτές και υπάρχουν σήμερα μεν πιέσεις ε, στις παράκτιες περιοχές, πολύ σημαντικές, που θα ήθελαν, όπως είπαν και εσείς, είπατε και εσείς, να αντικατασταθεί η θεοκαλλιέργεια ε, και τα οστρακοειδή και όλα αυτά που καλλιεργούνται για να αντικατασταθούν από άλλες δραστηριότητες. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να ε, ευαισθητοποιηθούν ε, οι δημόσιοι φορείς αλλά κυρίως το ευρύ κοινό και να γνωρίζει ποια είναι η κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα της ε, μιας δραστηριότητας όπως για παράδειγμα της καλλιέργειας οστρακοειδών ε, στο συγκεκριμένο κόλπο ή ηχθοκαλλιέργειας στη Βρετάνη και αλλού. Και μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που στόχο έχουν την ανάπτυξη ε, των ακτών στη Βρετάνη, οι τοπικές αρχές θέλησαν να αντιληφθεί και η τοπική κοινότητα τι συνέπειες υπάρχουν για αυτούς από τις αλλιευτικές ε, δραστηριότητες και την ηχθειοκαλλιέργεια. Αυτή τη στιγμή αφήκνονται νέε δραστηριότητε συνήθω, οι οποίε ε, φαίνονται πολλά υποσχόμενε αρχικώ. Μπορεί να επαληθευτεί, μπορεί και όχι, αλλά επειδή ακόμα δεν έχουν ε, δημιουργηθεί, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό με ε, βεβαιότητα, αλλά αρχίζει ο καθένας να είναι επιφυλακτικός απέναντι στις παραδοσιακές δραστηριότητες και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι ένας τρόπος για να αρχίσουμε να προστατεύουμε αυτές τις παραδοσιακές δραστηριότητες που είναι μεγάλη σημασία και ορισμένες φορές δεν έχουν και την θετική εικόνα που θα έπρεπε να έχουν. Υποτιμούνται οι κοινωνικο-οικονομικές συνέπειές τους και είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να προβάλλουμε μέσω αυτού του προγράμματος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κεντέλ θέλει να θέσει μια ερώτηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ουσιαστικά πέρασα όλη μου τη ζωή στη γέφυρα ενός σκάφους ως ε, αλλιεύς και ε, ελάχιστος είναι ο χρόνος ε, με τον οποίο ασχολούμαι με αυτές τις δραστηριότητες. Νομίζω ότι δεν ε, συνειδητοποιούμε απόλυτα κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη θέλουμε να αναπτύξουμε την ηχθειοκαλλιέργεια και δεν αντιλαμβανόμαστε τι φέρπει. Το ανέφερα ε, εντάχει. Τι χρειάζεται αυτός ο τομέας για να αναπτυχθεί, για να μπορεί ε, να ε, εκτρέφει σαρκοβόρα ψάρια. Χρειάζονται ζωοτροφές, ηχθιάλευρα, ε, τα οποία προέρχονται από ε, ψάρια ελεύθερα, μικρού μεγέθους ή μικρά ψάρια τα οποία χρησιμεύουν ως τροφή για μεγαλύτερα ψάρια και ε, είπα και μια ευχή την οποία ίσως δεν προσέξατε αυτό θα έπρεπε να συνεισφέρει στην ε, βιωσιμότητα αυτής της δραστηριότητας, δηλαδή ε, το να ε, χρησιμοποιούνται μικρά ψάρια για την παραγωγή χθιαλεύρων. Αυτοί οι χώροι τους οποίους εγώ αποκαλώ υγρότοπους είναι πολύ σημαντικοί διότι η παγκόσμια χρήση και επιμένω οδήγησε σε εισαγωγές ψαριών από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα και εξαγωγή κοινωνικο-οικονομικής μιζέριας, διότι αυτά τα προϊόντα που εισάγουμε δεν παράγονται με τις ίδιες προϋποθέσεις που επιβάλλουμε εμείς, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και οικολογικά προβλήματα, όπως διευκρίνησε ο κύριος ε, Σάντες. Και υπάρχουν λοιπόν ε, κάποια προβλήματα τα οποία είναι και αυτά παγκοσμιοποιημένα. Δεν παγκοσμιοποιούνται μόνο οι αγορές. Και κάτι ακόμα, το οποίο αφορά την Ευρώπη πιο συγκεκριμένα. Σε μια έκθεση του 2006 που διάβασα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, η κυρία Μακλέιτ, που ήταν τότε εκτελεστική διευθύντρια, έλεγε ότι Υπάρχουν παραδείγματα τα οποία αποδεικνύουν ότι ε, η περιβαλλοντική φορολογία μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση των εσόδων, στην οικονομία, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ε, ταυτόχρονα ε, προστατεύοντας και το περιβάλλον. Κάπου λοιπόν θα πρέπει να μελετήσουμε ως πιθανή ευκαιρία τη δυνατότητα να υπάρχει περιβαλλοντική φορολογία, η οποία όμως θα προέρχεται όχι ως κύρωση, αλλά ως προσαρμογή που θα μας επιτρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των διαφόρων τομέων. Διότι μέσω της ανάπτυξης του οικονομικού πλούτου, για παράδειγμα, που προέρχεται από τις ε, θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπάρχουν τεράστιες επενδύσεις και ε, υπάρχει και η ανησυχία και θα πρέπει το σύστημα αυτό να μπορεί να ε, χρηματοδοτωθεί και μέσω φορολογικής, ε, φορολογίας των περιβάλλων και ταυτόχρονα Ε, διατηρώντας την αλληλεία, ε, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει και αυτή σε αύξηση εισοδημάτων και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι για τα, τον τρόπο με τον οποίο θρέφονται τα σαρκοβόρα ψάρια, πραγματικά εγώ πρέπει να σας πω ότι ε, είμαι σε δυσάρεστη θέση. Εμείς πάντα ε, στη θάλασσα, και δεν υπήρχαν τότε ε, κίνητρα για καλύτερη συμπεριφορά, διότι αυτό είναι ο πόλεμος της θάλασσας, ε, η καλύτερη συμπεριφορά που θα πρέπει να οδηγήσει σε καλύτερες πρακτικές. Και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να το μελετήσουμε κάπου. Ευχαριστώ. να έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ και σας. η άποψή σας για την υδατοκαλλιέργεια είναι πολύ σημαντική. Και θα ήθελα να πω ότι ε, συμφωνούμε εμείς ε, με αυτό που είπατε όσον αφορά την εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλοι καλές πρακτικές. Ό,τι έγινε έγινε. Το παρόν είναι μια διαφορετική κατάσταση και ελπίζουμε ότι το μέλλον θα είναι ακόμα καλύτερο από το παρόν. Και νομίζω ότι διδαχθήκαμε από τα μαθήματα του παρελθόντων. Παραδείγματο χάρη, όσον αφορά την ηχθειοκαλλιέργεια, γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη σε κάποιες περιοχές, ε, ε, κυρίω στην Ασία και όχι τόσο στην Ευρώπη. και ξέρουμε ότι θα υπάρξουν ε, έντονες επενδύσεις ε, στην υδατοκαλλιέργεια. Υπάρχουν όλες οι ενδείξεις ε, προς αυτή την κατεύθυνση για το διάστημα 2014-2020 και εγώ πραγματικά ελπίζω ότι αυτή η ανάπτυξη της ηχθειοκαλλιέργειας στην Ευρώπη θα γίνει με βάση τα διδάγματα τα οποία έχουμε αντλήσει από αλλού. Ε, όσον αφορά όλα όσα ε, θίξατε εδώ ε, την παρουσίασή σας, συμφωνώ. Ο πρόεδρος, ο κύριος Στίβενσον, θα ήθελε να πει ένα-δυο πράγματα για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά ήθελα να αναφερθώ σε κάποια πράγματα που είπε ο κύριος Καντέλος, όσον αφορά τα αλευρά. Είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε συνεχώς ε, στην Επιτροπή Αλίας. Υπάρχει πολλή ανησυχία ότι η χρήση ηχθιάλευρων και ηχθιελαίων ε, δεν είναι βιώσιμη. Έχουμε στείλει στο παρελθόν ε, αντιπροσωπείες στη Χιλή και στο Περού για να εξετάσουν τη βιωσιμότητα του σχετικού τομέα. Και πρέπει να σας πω ότι και για τους κολλιούς και για τις ε, αντζούγες ε, έχει ε, αναγνωριστεί η βιωσιμότητα και στη Χιλή και στο Περού. Ωστόσο, πριν 10 χρόνια η αναλογία ηχθιάλευρου και ηχθιελαίων που δίνονταν σε ψάρια ηχθειοκαλλιέργεια. ήταν ε, κατά μέσο όρο 7 ε, με 10 κιλά για παραγωγή ενό κιλού ε, ψαριού για πώληση. Τώρα ε, ο τομέας έχει βελτιώσει τις τεχνικές του και ε, το, η ποσότητα αυτή είναι 2 ε, κιλά σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και 1,5 κιλό ανά παραγόμενου κιλού. σε κάποιες περιπτώσεις τα ε, ψάρια της ηχθειοκαλλιέργειας ε, ε, τρώνε τελικά λιγότερο ηχθιάλευρο και ηχθιέλαιο από ό,τι θα ελάμβαναν στο, εάν, εάν ζούσαν στη θάλασσα, εάν ήταν Εάν ήταν ψάρια θαλάσσιος και όχι ηχθειοκαλλιέργειας. Και χθε το βράδυ είχαμε τι διαπραγματεύσει για την μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, κάτι που περιλάμβανε και το θέμα των απορρίψεων. Η αλληλείς της Ευρώπης ε, ποτέ ε, δεν δέχτηκαν, ποτέ δεν τους άρεσε αυτό το μέτρο που τους επιβλήθηκε. Η ε, Κομισιόν υπολόγισε ότι 1,7 εκατομμύρια τόνοι απορρίπτονταν ανά χρόνο στα ευρωπαϊκά ύδατα και ο πυρήνας της μεταρρύθμισής μας όσον αφορά την απαγόρευση των απορρίψεων στόχο έχει να αφήνουμε τα ε, ψάρια στη θάλασσα, να εφαρμοστούν τεχνικά μέτρα ώστε να αποφεύγεται η αλία των ψαρών αυτών. Ε, ωστόσο, τα μικρά αυτά ψάρια ή τα ψάρια που ε, ξεπερνούν τις ποσοστώσεις που συνεχίζουν να εκφορτώνονται σύμφωνα με την απαγόρευση απορρίψεων θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηχθιάλευρων και ελπίζουμε ότι έτσι θα μειωθεί το κόστος ηχθιάλευρων και ηχθιελαίων, κάτι που θα κάνει πιο ανταγωνιστικό τον, ε, το, ε, θα κάνει πιο ανταγωνιστική την ηχθιακαλλιέργειά μας. Ε, το άλλο που θα ήθελα να πω ήταν ότι αρκετοί από τους ομιλητές σήμερα μίλησαν για το 65% των, εισαγωγών, των εισαγόμενων ψαριών από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου τα πρότυπα είναι χαμηλά, τα κοινωνικο-οικονομικά πρότυπα επίσης εγώ παλιά ήμουνα σημαντικός ε, επικριτής ε, του ψαριού Παγκάσιους ε, που, ερχόταν, που προέρχεται από το Βιετνάμ. Η Κομισιόν λόγω έλλειψης δυναμικού έστελνε επιθεωρητές μόνο μια φορά, το χρόνο, μια φορά στα δύο-τρία χρόνια για να επιθεωρήσουν τις εγκαταστάσεις στον στο Βιετνάμ ε, και εμείς είπαμε ότι αυτό δεν αρκεί. Ε, ακούμε ότι το ψάρι αυτό είναι πολύ χαμηλής ποιότητας, ε, παράγεται σε υποσυνθήκες κακής υγιεινής. Και πήγα κι εγώ ο ίδιος στο Νόμιλο Βενχόγκ, όπου 6.000 γυναίκες εργάζονται στο πιο καθαρό δυνατό περιβάλλον, διότι είπαν ότι Δεν μας πειράζει που έρχονται οι επιθεωρητές σας σε μόνο πέντε χρόνια. Οι Κάρφουρ, οι Τέσκο, οι Άστα μας επιθεωρούν κάθε χρόνο. Ακόμα και οι αρχές της Αμερικής, επειδή πολλούν, εξάγουν και εκεί τα ψάρια τους. Και πιστέψτε με, Έχω επισκεφτεί πολλές εγκαταστάσεις μεταποίησης στην Ευρώπη, αλλά αυτό που είδα ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Φυσικά είναι πολύ πιο χαμηλές οι αμοιβέ τους από τις δικές μας ε, και αυτό τους κάνει ανταγωνιστικούς. Ε, αλλά ζούμε σε, ε, στα πλαίσια μιας παγκόσμιας αγοράς Εάν λοιπόν ε, είμαστε υποχρεωμένοι να ε, καλύψουμε αυτό το κενό το 65% μπορούμε να το κάνουμε μόνο ε, πολλώντας ψάρια που έχουν παραχθεί με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα σε όλο τον κόσμο και θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά. Ποτέ δεν θα έχουμε συνθήκες ίσου ανταγωνισμού, δεν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά σας παρακαλώ μην νομίζετε ότι οι εισαγωγές αυτές είναι κακής ποιότητας και ότι παράγονται υπό συνθήκες κακής Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το πάνελ. Ε, έχουμε ακόμα χρόνο και μπορούμε να υποφεληθούμε από την παρουσία των προσκεκλημένων μας. Ε, και εγώ έχω κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με αυτά που είπατε. Δεν ε, μπορούμε... Να, δεν πρέπει να πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Να λέμε δηλαδή ότι όλα τα ε, ψάρια που εισάγονται είναι κακά, ε, αλλά εξίσου ακραίο θα ήταν να λέμε ότι όλα τα ε, ψάρια που εισάγονται είναι καλά. Είχαμε τώρα την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Ταϊλάνδη, που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας τόνου και ξέρω το 2012 Η αξία των εξαγωγών τόνου από την Ταϊλάνδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε λίγο. Ξέρετε όμως γιατί. Να το πω στα πορτογαλικά. Γιατί οι κονσέρβες ήταν ελαττωματικές. Ε, οι συσκευασίες εννοώ. Και χρειάστηκε να επιστραφούν στην Ταϊλάνδη. Το γεγονός αυτό ότι η ίδια η συσκευασία ε, ήταν αυτοματική, σημαίνει ότι και επηρεαζόταν και η ποιότητα του ψαριού. Χρειάζεται λοιπόν να διατηρήσουμε μια ισορροπία σε όλα αυτά. Το καλύτερο είναι να αναπτύξουμε τον αλευτικό τομέα και το τομέα της στην Ευρώπη. Uh, Θα ήθελα να τονίσω δύο ακόμα πράγματα που θεωρώ πολύ σημαντικά. Ξέρω ότι έχουμε ακόμα χρόνο. Δεν κλέβω λοιπόν χρόνο από το επόμενο πάνελ. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω μια άλλη ερώτηση προς τους ε, ομιλητές μας. Ο κύριος ε, Ρικάρτο ε, Σάντος μίλησε για την προστασία κάποιων συγκεκριμένων περιοχών. Και επίσης μας έδωσε ενδιαφέροντα παραδείγματα από τις Αζόρες, όπου υπάρχουν τέτοιες περιοχές. Οι αλληλείς συμφωνούν με την προστασία των περιοχών αυτών ε, και ε, την στηρίζουν. Εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο δεν θα πρέπει να υπάρχει αμφιβολία σχετικά με το ότι πρέπει να περιοριστεί η μεγάλη αλληλευτική προσπάθεια στις περιοχές αυτές. Ε, και ε, κάποτε πρότεινα στο Κοινοβούλιο η, τα ευάλωτα αυτά θαλάσσια οικοσυστήματα να προστατεύονται από τους μεγάλους στόλους και οι αλλιευτικές δραστηριότητες σε αυτές τις περιοχές να περιορίζεται σε αλία μικρής κλίμακας. Να επιτρέπεται στον περιφερειακό στόλο μόνο και να μην είναι ανοιχτή για όλο τον ευρωπαϊκό στόλο που είναι πολύ μεγαλύτερος ε, από τον ε, τοπικό στόλο. Εξεπλάγιν που η πλειοψηφία της σοσιαλιστικής ομάδας ε, δεν στήριξαν την ομάδα αυτή. Ούτε καν οι πράσινοι δεν συμφώνησαν. Μερικές φορές λοιπόν πραγματικά καταλάβ... Ε, δυσκολεύομαι να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει εδώ, διότι έχουμε αυτές τις ευάλωτες θαλάσσιες περιοχές οι οποίες προστατεύονται για ε, περιβαλλοντικούς λόγους. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο συνεπείς όσον αφορά το τι θεωρούμε σημαντικό. Και θα ήθελα να ζητήσω από τον δόκτωρο Ρικάρδο Σερασάντος ε, να μας ε, μιλήσει περισσότερο, ε, περισσότερο σχετικά με τη σημασία της προστασίας των υφάλων γύρω από τις Αζόρες. Μιλάμε για το κέντρο του Ατλαντικού ωκεανού. Είναι δηλαδή σημαντικά αυτά, όχι μόνο για τα νησιά αυτά, αλλά για το σύνολο των οικοσυστημάτων στο βαρά του Ατλαντικού. Θα παρακαλούσα λοιπόν να αναφερθείτε σε αυτό και και όσον αφορά την παρουσίαση του κυρίου ε, Κάρλε Κίντ, ήταν πολύ σημαντικό που μιλήσατε ε, όχι μόνο για, το, για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις αλλά και τις ε, κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις. Όλοι μας εδώ στο Κιλεβόνιο γνωρίζουμε ότι και εγώ ως για την πράσινη βίβλο για την μεταρρύθμιση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής επέμεινα και επιμένουμε στην ισορροπία μεταξύ των τριών πυλώνων. Εγώ πάντοτε λέω ότι δεν είναι δυνατόν να προβάλλουμε μόνο τον περιβαλλοντικό πυλώνα λέγοντας ότι θα ε, αναλάβουμε να επιλύσουμε όλα τα περιβαλλοντικά και οικολογικά προβλήματα και αργότερα θα επιληφθούμε των υπόλοιπων κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων. Η ζωή δεν λειτουργεί έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, που εξαρτώνται από την δραστηριότητά τους στη θάλασσα και ιδιαίτερα από την αλία. Συνεπώς ε, ήταν πολύ ενδιαφέρον που μιλήσατε κι εσείς για τους τρεις ακριβώς πυλώνες. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για την ανάγκη και τα ε, πλέον εκτίματα μιας καλής ισορροπίας μεταξύ αυτών των τριών πυλώνων. Ρικάρδο. Ε, ε, Το 2007 δημοσίευσαμε ένα βιβλίο για, την αλία σε ε, υποθαλάσσια όρη ε, έδειχνε ότι αυτό το είδος της αλίας από τη φύση του ε, είναι διάσπαρτο, είναι σε μεγάλες γεωγραφικές ζώνες. Η παραδοσιακή αλία και αλία μικρής κλίμακας είναι πιο βιώσιμη και καταλαμβάνουν όλη την κλίμακα αλλιές σε μια ζώνη, σε μια περιοχή. Ε, καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα, απασχολούν περισσότερο προσωπικό και είναι πιο αποδοτικές. Συνεπώς η αλία μικρής κλίμακας και η παράκτη αλία ε, έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει αντιληφθεί. Γι' αυτό το λόγο και ξέδωσε το ψήφισμα του 2005. Έτσι ώστε να μειωθεί η αλία σε υποθαλάσσια βουνά. όρι. Κρίστοφερ Φαμ μίλησε για το υποθαλάσσιο της Κοντόρας της Αζόρες. Ε, η, γίνεται, η αλία εκεί γίνεται με ε, σταθερά, σταθερές καθέ, καθετές, ε, κα, ε, βυθού αντίθετα είναι καλύτερο η, να γίνεται με χειροκίνητες καθετές ε, που είναι κάτι πολύ πιο οικολογικό διότι δεν καταστρέφουν το θαλάσσιο περιβάλλον και αυτές γίνονται από τις ε, αποτελευτικά ε, μικρής κλίμακας και την, τους παράκτιους αλίες. Euh, euh, ναι, κυρία θα πρέπει να σκεφτούμε τις τρεις βασικές ε, πτυχές της ε, ανάπτυξης, ε, της βιώσιμης ανάπτυξης, κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στις παράκτητες περιοχές στη Βρετάνη, τις οποίες γνωρίζω λίγο καλύτερα. Δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής χωρίς να λάβουμε υπόψη και τους τρεις πυλώνες. Σήμερα Εάν ε, ε, καταφέρουμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό, κάτι το οποίο επιθυμούν αυτές οι περιοχές, διότι και αυτό είναι παράγον ανάπτυξης, ε, ξέρουμε πόσο θα περιοριστούν άλλες παραδοσιακές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα λιαυτικές δραστηριότητες. Είναι αλήθεια ότι όταν δημιουργηθεί ένας κοινωνικός και οικονομικός ιστός μόνιμος, ε, οι αλλιευτικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες μεταποίησης των αλλιευτικών προϊόντων δημιουργούν και μόνιμες δομές ε, όπως παραδείγματο χάρη ε, το εμπόριο σε μια πόλη, σε μια κοινότητα, διότι ε, ζουν από τις ελευτικές δραστηριότητες και από εκεί και πέρα υπάρχει και όφελος για τον τουρισμό. Ο τουρισμός ορισμένες φορές ε, προέρχεται ως δέλεαρ των αλληλευτικών δραστηριοτήτων. Όταν κάποιος είναι τουρίστας, ε, σας το λέω έτσι λίγο και, ε, ανόητο ίσως, αλλά χαίρεται να βλέπει κάποιον να ψαρεύει. Υπάρχει λοιπόν στενή σχέση μεταξύ της κοινωνικής ζωής, κοινωνικής ανάπτυξης και εδαφικής συνοχής, θα τα βάλω και αυτά μαζί, και της οικονομικής ανάπτυξης. Και η ανάγκη να έχουμε φυσικά και μια περιβαλλοντική διάσταξη είναι εξίσου σημαντική για να σεβόμαστε του πόρου μα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αλλιεύσο ο οποίο δεν είναι απόλυτα πεπισμένο ότι το πρώτο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι η κατάλληλη διαχείριση των πόρων, ευφυή συλλογική διαχείριση των πόρων αυτών που ταυτόχρονα θα είναι και μια ευφυή συλλογική διαχείριση τη ποιότητα του περιβάλλοντο το οποίο αναπτύσσονται ...αυτή οι πόροι. Και για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, ο, για να επανέλθω στον τουρισμό, ο τουρίστας ε, ευχαρίστως ε, θα απολαύσει μια υγιή περιοχή όταν έρχεται να κάνει μια βόλτα σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Και μπορεί βέβαια να κάνουν και προβλέψεις αποκάλυψης, αλλά εάν ε, διανοηθεί κανείς κάποιες περιοχές της Βρετάνης χωρίς αλληλεία, ε, μπορεί να χάσουμε και όλες τις υπόλοιπες, διότι η αλληλεία επιτρέπει να υπάρχει μια καθημερινότητα η οποία δίνει ε, και ε, άλλες εργασίες και γεννά και άλλες εργασίες και αυτό είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ. Ήρθε η στιγμή τώρα για το επόμενο πάνελ. Αλλά η Ντολόρες ε, θέλει το λόγο. Αν είναι δυνατόν να είστε σύντομοι. Ναι, ευχαριστώ. Καταρχάς ζητώ συγγνώμη γιατί ήρθα λίγο καθυστερημένη, αλλά έπρεπε να ε, ε, πάω και σε μια άλλη επιτροπή. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η αξιολόγηση που έκαναν οι δύο πυρογνώμονες και νομίζω ότι συμπίπτει και με την δική μου τη θέση, την οποία προασπίζομαι, και εν γέννη με τη θέση των χωρών της Νότιας Ευρώπης. Αν θέλουμε να έχουμε μια αλληλευτική πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη της κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές, ε, τότε αναφερόμαστε σίγουρα στην αλληλεία μικρής κλίμακας. Και για μένα είναι θλιβερό το γεγονός ότι τελικώς αυτή τη μεταρρύθμιση που γίνεται μόνο ε, κάθε 10 χρόνια, η αλληλεία μικρής κλίμακας είναι ο μεγάλος ξεχασμένος. Ε, η συγκεκριμένη αλληλεία όχι μόνο δημιουργεί θέσεις εργασίας, αλλά ε, και προστατεύει τη θάλασσα περισσότερο και μπορεί να αποτελέσει και δέλεαρ για βιώσιμο τουρισμό. Υπάρχουν τεράστιες περιοχές, χωριά, πόλεις που ζουν από αυτή τη δραστηριότητα και με τη νέα πολιτική ε, δεν νομίζω ότι θα χάσουμε για πάντα τις απορρίψεις, αλλά θα αντικατασταθούν οι απορρίψεις από μια αγορά ηχθιαλεύρων που θα είναι εις βάρος ε, της αλίας μικρής κλίμακας. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση κατά της υδατοκαλλιέργειας, αλλά πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη ισορροπία. Ο καταναλωτής ε, θα έχει να επιλέξει ανάμεσα σε ένα προϊόν της θάλασσας και ένα προϊόν το οποίο θα έχει παρασκευαστεί ε, σε ένα κλειστό χώρο με διάφορες εγγύσεις. Ε, εγώ επιμένω ότι θα είναι δύσκολο, όχι σε οικονομικούς όρους, γιατί είναι βιώσιμο, αλλά σε κοινωνικούς όρους, όταν δεν γνωρίζουμε πού αλλιεύουμε, πώς παράγονται ε, ή πώς μεταποιούνται όταν μιλάμε για μεταποιημένα προϊόντα. Ε, αναφερθήκατε σε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, τις προστατευόμενες περιοχές. Και όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Η ερώτηση λοιπόν για τον κύριο Σάντος είναι, αν δεν κάνω λάθος, ε, στην Ισπανία αυτή τη στιγμή ε, προωθείται ένα ευρύτερο δίκτυο προστατευμένων περιοχών. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για το τι συμβαίνει στη χώρα μου. Εγώ είμαι από την Ισπανία. Ρικάρτο, ε, θα μπορούσε να απαντήσει σε, σε, εν συντομία, βέβαια, για να μην κλέβουμε χρόνο από το επόμενο πάνελ. Ε, δεν κατάλαβα πολύ καλά την ερώτηση. Σε ό,τι αφορά την Ισπανία, τι γίνεται με το δίκτυο των προστατευόμενων ε, περιοχών, ξέρεις τι εξελίξεις υπάρχουν στην Ισπανία. Ναι, έχει προχωρήσει πολύ πιστεύω. Το project του FP6 Ε, με επικεφαλή στην Μούρθια. Ε, λαμβάνει χώρα στις προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου. Και πιο πρόσφατα οι προτάσεις για την ΟΣΠΑΡ, την προστασία των υποθαλάσσιων ωραίων και κάποιες προτάσεις ακόμα από Ισπανούς συναδέλφους για την δημιουργία προστατευόμενων ζώνων στο νότιο Ατλαντικό, ε, αλευτικές ζώνες ε, ε ισπανικών σκαφών συγκεκριμένα, νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν πως η Ισπανία κάνει σημαντικά βήματα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πολιτική υποστήριξη για τα ε, επιτεύγματα. Ήταν χαρά μου να είμαι πρόεδρος σε αυτό το πάνελ και τώρα είναι σειρά της συναδέφου να παρουσιάσει το επόμενο πάνελ. Επιτρέψτε μου πρώτα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Πατράου ε, που προέδρευσε εξαιρετικά στο δεύτερο πάνελ και να καλωσορίσω την κυρία Μάισνερ που θα προεδρεύσει στο επόμενο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσθέσω άλλη μία γλώσσα. Θα μιλήσω λοιπόν πρώτα στα γερμανικά και μετά στα αγγλικά. Προχωράμε τώρα στο τρίτο πάνελ. Και να πω καταρχήν ότι λυπάμαι πάρα πολύ που δεν ήμουν παρούσα στη συζήτηση των άλλων δύο, διότι ζήτησα να οργανωθεί αυτή η ακρόαση, διότι πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό η Επιτροπή Αλληλείας ε, να έχει μια πιο ε, ευρεία εικόνα της θάλασσας. Ήμουνα όμως συντονίστρια σε μια μακρά ψηφοφορία, δεν μπόρεσα να είμαι παρούσα. Ο ο βοηθό μου όμω είναι εδώ και νομίζω θα με ενημερώσει σχετικά με το όσα είπαν η Ιζαμπέλ και η Μαρία, διότι είναι πολύ σημαντικά αυτά. Και όσα είπαν φυσικά και οι άλλοι ομιλητέ. Ε, ε, γιατί λοιπόν με ενδιαφέρει αυτό το θέμα αυτό. Ε, δεν συμμετέχω μόνο στην ε, Επιτροπή Αλίας, ε, συμμετέχω και στην Επιτροπή μεταφορών ε, και ήμουνα εισηγήτρια για ε, την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική που ξεκίνησε το 2007 και είναι πάρα πολύ σημαντικό Όλε τι δραστηριότητε τη θάλασσα να τις ε, εξετάσουμε μαζί ώστε να έχουμε βιώσιμη εκμετάλλευση και χρήση της θάλασσα. Μπορεί αυτό να μην είναι πάρα πολύ γνωστό. Η Επίτροπος είναι η αρμόδια για η Επίτροπος είναι αρμόδια για θέματα ε, ε, αλληλείας ε, και θαλάσσης γενικά, αλλά εδώ πέρα επί της ουσίας αρμόδια για τις ολοκληρωμένες θάλασσες μεταφορές είναι η Επιτροπή Μεταφορών. Ξέρετε ότι ο κόσμος έχει 70% θάλασσα και 30% γη, είναι γνωστό αυτό, αλλά το επαναλαμβάνω και αυξάνεται ο πληθυσμός της γης και γι' αυτό χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο και τη θάλασσα. Ε, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, την ε, ευαισθησία της θάλασσας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε μια λογική ανάπτυξη. Ακούσαμε διάφορα. Ξέρω ότι τα άλλα πάνελ αναφέρθηκαν σε διάφορες περιφέρειες, τη Βρετάνη, τις Αζόρες, την Ισπανία, τον Νότο της Ευρώπης. Εγώ θα προσθέσω μια άλλη πτυχή της ε, Βόρειας ε, Ευρώπης, ε, Γερμανίδα είμαι και μάλιστα οι βοηθοί μου προέρχονται από την Γερμανία και, την, και τις κάτω χώρες αντίστοιχα. Πρόκειται λοιπόν για μια άλλη πτυχή, οι ομιλητές μου, συγγνώμη, και θα... Το θέμα είναι η παράλληλη ανάπτυξη της αλίας που είναι πολύ παλιά δραστηριότητα με, ε, με την ε, ηχθειοκαλλιέργεια, με τις θαλάσσιες μεταφορές, με τις παράκτιες τεχνολογίες ε, και όσον αφορά την εξόριξη πετρελαίου και αερίου, αλλά και όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε περισσότερες εξορίξεις από τη θάλασσα ε, και άλλωστε και ο κόσμο ε, πολύ ευχαρίστω περνάει τι διακοπέ του στην ακτή. Χρειαζόμαστε λοιπόν και βιώσιμο τουρισμό. Κλείνοντα λοιπόν την εισαγωγή μου, θα ήθελα να πω ότι στην περιφέρειά μου, στην ε, Βόρεια Θάλασσα, έχουμε εκεί μια, ένα μοναδικό οικοσύστημα ε, στις κάτω χώρες και στην Γερμανία, στις ακτές εκεί στα ε, ε, ε, λείπει η Δανία από την ζώνη αυτή, αλλά ελπίζουμε αυτό να διορθωθεί. Πρόκειται λοιπόν για μια περιοχή όπου αναπτύσσεται ο τουρισμός και γίνονται όμως και θαλάσσιες μεταφορές, υπάρχουν παράκτιες εγκαταστάσεις, αλληλεία. Στην περιοχή αυτή λοιπόν ε, ε, συνδυάζονται όλες οι δραστηριότητες. Χαίρομαι λοιπόν που είμαι η συγγήτρια του Κοινοβουλίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ε, ώστε να μπορέσουμε να, αναπτύξουμε ε, περισσότερο το θέμα. Ε, τελευταία μου παρατήρηση, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα ως εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου στην Μάλτα για την Ευρωπαϊκή Μέρα Θαλάσσης και ένιωσα εκεί πόσο ε, Σημαντικό είναι ο χωροταξικό σχεδιασμό και η διαχείριση των ακτών για όλους τους φορείς στον τομέα αυτών. Ε, υπήρξε πολύ έντονο ενδιαφέρον ε, και πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι η η Γερμανίδα Καγκελάριος Μέρκελ, που δεν είναι άγνωστη, ρωτήθηκε πρόσφατα ε, αν δεν έπρεπε συνέχεια να λύνεται την κρίση στην Ευρώπη ως ε, πολιτική για το μέλλον, με τι θα ασχολιόσασταν. Ε, και εκείνη απάντησε με την θαλάσσια πολιτική. Είναι άλλωστε επιστήμον και όπως και άλλη πολιτική γνωρίζει πολύ καλά πόσο σημαντικός είναι ο τομέας αυτός. Περνώ λοιπόν τώρα στους δύο ομιλητές μου. Έχω καλέσει ε, δύο ομιλητές. Ε, θα μιλήσω αγγλικά ε, η πρώτη ομιλήτρια είναι η κυρία Βανέσα Στέλσεν ε, Βρίσκεται μπροστά από το λάπτοπ ε, ήδη. Είναι επιστήμον στο Ινστιτούτο Αλίας στο Αμβούργο και ασχολείται με τη διαχείριση της θάλασσας και το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς και την επίλυση διαφορών ανάμεσα στους αλληλείς και άλλους χρήστες της θάλασσας. Είναι η πρώτη μου ομιλήτρια. Να παρουσιάσω ήδη τον δεύτερο ομιλητή μου, βρίσκεται εδώ στη μέση της αίθουσας ε, είναι ο Ντάβιντ Γκόλσπορο. Σωστά το προέφερα, δεν είμαι σίγουρη. Λίγο πολύ καλά. Θα με διορθώσετε. David Γκόλσπορο; Είναι ερευνητής και λέκτορας ε, στο Πανεπιστήμιο Wageningen. Στις κάτω χώρες, όπως σας είπα. Είναι πανεπιστήμιο με πολύ καλή φήμη όσον αφορά την ε, θαλάσσια οικολογία. Έχει Ινστιτούτο ε, Θαλασσίων ε, Ερευνών, η ΜΑΡΕΣ ίσως να το γνωρίζετε. Ε, και έχει κέντρο θαλάσσιας πολιτικής το πανεπιστήμιο αυτό. Ασχολείται με το πρόγραμμα μάσπνος το οποίο επιδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, έχει ασχοληθεί με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ιδιαίτερα στη Βόρεια Θάλασσα. Οι δύο ερευνητέ αυτοί λοιπόν μπορούν να συμπληρώσουν την εικόνα που έχουμε λάβει μέχρι τώρα, εξηγώντα μα πρακτικέ εφαρμογέ σχετικά με τον ε, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Αυτή ήταν η εισαγωγή μου λοιπόν. Ε, τους δίνω το λόγο, παρακαλώ. All right. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Θα ήθελα να σας δείξω κάποια αποτελέσματα κάποιων μελετών που εξετάζουν τα αποτελέσματα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στα αλλιεύματα και στην αλληλεία στη Βόρεια Θάλασσα. Η Βόρεια Θάλασσα ε, είναι πολύ ιδιαίτερη. Βλέπετε εδώ πώς ε, γίνεται η διανομή στο χώρο. Έχουμε δραστηριότητες, εξόριξη πετρελαίου και φυσικού αερίου και ε, εδώ με μπλε χρώμα έχουμε αυτές τις δραστηριότητες, έχουμε επίσης αλληλεία και με πράσινο έχουμε κάποιες ε, περιοχές ε, προστατευόμενες καθώς επίσης περιοχές οι οποίες βρίσκονται είτε σε παράκτιες περιοχές είτε κοντά στις ακτές. Ε, υπάρχει και μεγάλος βαθμός αλληλοεπικάλυψης μεταξύ των δραστηριοτήτων και αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Ε, στην ε, Βόρεια Θάλασσα ο θαλάσσιος χωροταξιακός ε, σχεδιασμός ε, είχε ως βασικό παράδειγμα την εξόριξη πετρελαίου και το φυσικό αέριο και επομένως αρκετές χώρες θεώρησαν ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει κατάλληλος χωροταξικός σχεδιασμός. Το βασικό πρόβλημα είναι η ναυτιλία και τα ελλικά πάρκα και επίσης προστατευόμενες περιοχές και αλία. Δεν υπάρχει κάποια περίπτωση στην οποία να περιλαμβάνεται και η αλληλεία σε κάποιες περιοχές ε, ως προτεραιότητα. Θα ε, μιλήσω καταρχάς ε, για τη γερμανική εμπειρία και εξετάσαμε λίγο τι συνέπειες μπορεί να έχουν οι υδατοκαλλιέργειες. Στην αριστερή στην αριστερή πλευρά έχετε το γερμανικό χωροταξικό σχέδιο και θα ήθελα να σας αναφέρω τις κόκκινες περιοχές που είναι οι περιοχές ε, προτεραιότητας για την ανάπτυξη των αιωλικών πάρκων. Ε, Απ' την άλλη πλευρά βλέπετε τις ε, εγκεκριμένες ε, περιοχές όπου έχουμε αιωλικά πάρκα και επίσης υπάρχουν και κάποιες αιτήσει για ε, αιωλικά πάρκα παράκτια, τα οποία είναι υπό επεξεργασία αυτή τη στιγμή. Και θα πρέπει να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει συγκεκριμένο ε, σχέδιο χωροταξικό ε, για τη Γερμανία, εξακολουθούν να επεκτείνονται κάποιες ανθρώπινες δραστηριότητες και υπάρχουν κάποια αβεβαιότητα γιατί δεν ξέρουμε τι χωροταξικό σχεδιασμό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην γερμανική ζώνη αποκλειστικής εκμετάλλευσης και κοιτάμε να δούμε τι συνέπειες υπάρχουν για το περιβάλλον και άλλες χρήσεις ε, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Εξετάσαμε τις βασικές ανθρώπινες δραστηριότητες ε, στην γερμανική περιοχή και ε, χρησιμοποίησαμε τις πληροφορίες αυτές και εφαρμόσαμε στη συνέχεια και κάποιες δυνατότητες να υπάρχουν αντίθετες συνέπειες. Υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες οι οποίες αποκλείουν η μία την άλλη ή θα μπορούσαν να συνεπάρξουν σε μια περιοχή. Με βάση αυτό λοιπόν ετοιμάσαμε μια σειρά από χάρτες όπου βλέπουμε τομεί στους οποίους ε, μπορεί να υπάρχει δυνατότητα αντιθέσεων. Έχουμε λοιπόν ένα χάρτη στον οποίο έχουμε πολλές μαύρες περιοχές που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες εκεί οι οποίες αποκλείουν η μία την άλλη και αυτό εντείνεται και από την παρουσία διεθνών αλληλευτικών δραστηριοτήτων αλλά και προστατευόμενων περιοχών, γι' αυτό ε, ε καθώς επίσης συγγνώμη, και κάποιων ήδη εγκεκριμένων περιοχών όπου υπάρχουν αεολικά πάρκα. Πρέπει λοιπόν να δούμε ε, τι χρήσεις υπάρχουν, αλλά πρέπει να δούμε και τι συνέπειες έχουμε και για τους πόρους και για την αλληλεία ε, με βάση αυτή τη χρήση των πόρων. στόχος μας ήταν να προβλέψουμε τι συνέπειες θα έχουν τα μέτρα που λάβαμε και αν μπορούμε να έχουμε για παράδειγμα ε, πλήρη ανάπτυξη παράκτειων αιωλικών πάρκων. Κοιτάξαμε να δούμε τι συνέπειες θα έχουμε και χρησιμοποίησαμε και επιστημονικά δεδομένα για να ετοιμάσουμε μοντέλα παραγωγής. Ε, αυτά τα έχουμε στην αριστερή στήλη στις διαφάνειες και με σκούρο πορτοκαλί ε, είναι οι τομείς στους οποίους περιμένουμε αύξηση της βιομάζας και στη δεξιά στήλη βλέπετε ε, μία προσέγγιση όπου χρησιμοποίησαμε ε, στατιστικά δεδομένα αλληλείας, όπως ε, για παράδειγμα εκφορτώσεις, στοιχεία των μητρών του πλοίου και ετοιμάσαμε χάρτες για τα εισοδήματα που έχουμε, για παράδειγμα, στην γλώσσα, με την αλληλεία γλώσσας. Αυτά όλα πρέπει να τα εξετάσουμε όταν ε, ε, έχουμε το ψήφισμα για το χωροταξικό σχεδιασμό. Λαμβάνουμε υπόψη και τι γίνεται και με τα αεολικά πάρκα και κοιτάμε ε, τι μπορούμε να κάνουμε. Άλλωστε σε κάποιες περιοχές στις οποίες υπάρχει άνεμος δεν υπάρχει αλληλεία. Χρησιμοποίησαμε λοιπόν κάποιους κανόνες για να δούμε πού ε, μπορούμε να έχουμε κάποιες περιοχές στις οποίες θα έχουμε αποκλειστική δραστηριότητα και προσπαθήσαμε όλες αυτές τις πληροφορίες να τις συμπεριλάβουμε σε προηγμένα στατιστικά μοντέλα για να μπορέσουμε για παράδειγμα να ε, προβλέψουμε την ε, παρούσα κατάσταση των συνολικών αλευμάτων γλώσσες και να έχουμε και στην τρίτη ε, διαφάνεια, στην τρίτη χαρτογράφηση, τις προβλέψεις για τα συνολικά αλλιεύματα με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε αυτή τη μετατόπιση και τη συγκεκριμένη κατανομή των πόρων μας. Δύο στοιχεία θα ήθελα να αναφέρω εδώ. Υπάρχουν κάποια μοντέλα τα οποία μας δίνουν κάποιες προβλέψεις ε, για την πιθανή κατανομή των αλλιευμάτων, αλλά υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα με όλες αυτές τις ε, μεθόδους, διότι ακόμα δεν έχουν κατασκευαστεί τα αιωλικά πάρκα, έχουμε εγκρίνει κάποιες αιτήσει και επομένως ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο μεθόδους ανάλυσης κινδύνου με προβλέψεις και πρέπει όμως να τις λάβουμε και αυτές οι υπόψεις μας, αλλά υπάρχει και μεγάλη αβεβαιότητα ε, και για τα διάφορα ε, εναλλακτικά σενάρια για μετατόπιση και τι γίνεται όταν έχουμε για παράδειγμα αιωλικά πάρκα, τι βιολογικές συνέπειες υπάρχουν, τι ωφέλη και ούτω καθεξής. Όπως ακούσαμε ήδη και σήμερα το πρωί, η αλληλεία δεν σταματάει φυσικά στην ε, ε, ζώνη αποκλειστικής εκμετάλλευσης ε, στα χωρικά ύδατα, αλλά είναι διεθνή η δραστηριότητα. Γι' αυτό και ε, εδώ στη Βόρεια Θάλασσα ξέρουμε ότι δραστηριοποιείται και το Βέλγιο, η Δανία και οι κάτω χώρες. Με γκρι λοιπόν εδώ έχουμε όλε τι περιοχέ της τρει αυτέ χώρε όπου έχουν κατατεθεί αιτήσει για αεολικά πάρκα και υπάρχουν επίση και προστατευόμενε περιοχέ βάσει του Natura 2000. Εδώ υποθέτουμε ότι δεν θα υπάρχει αλληλεία στις ε, περιοχές που έχουμε ολικά πάρκα και ε, αποκλείονται και ε, βαθιά εργαλεία, εργαλεία που φτάνουν σε μεγάλο βάθος στις προστατευόμενες περιοχές από το Natura 2000. Κάνουμε και μία ανάλυση και βάσει των ε, ε, στοιχείων και των προβλέψουμε μέχρι και 90% των αλλιευτικών σκαφών των κάτω χωρών θα μπορούσαν ίσως να χάσουν παντελώς τη δραστηριότητά τους ε, επειδή θα κατασκευαστούν αυτά τα νέα αλλιευτικά, αιωλικά πάρκα. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάποιες μελέτες για να δούμε πώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν και την αλληλεία κάποια μέτρα για να συνοψίσω τώρα για τα βασικά μας αποτελέσματα, ε, αναμένουμε ότι θα υπάρξουν αντιθέσεις και διαφορές ε, από την ε, αλλαγή της χρήσης και την αύξηση κάποιων ε, δραστηριοτήτων και πρέπει να σας πω ότι θα υπάρχουν συνέπειες και σε ανθρώπινο και σε βιολογικό επίπεδο. Ε, όπως σας είπα όμως σε κάποια στοιχεία έχουμε πολύ περιορισμένες πληροφορίες γιατί δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν ε, τα αλλιευτικά σκάφη ε, σε κάποιες περιοχές που θα κλείσει και θα απαγορευτεί ε, η αλληλεία και δεν ξέρουμε και τι εμπορικά στοιχεία θα έχουμε για την αλληλεία. Και θα ήθελα να σας κάνω τρεις ε, παρατηρήσεις. Γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την εισαγωγή της αλληλείας στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Πρώτον, γιατί θα πρέπει να έχουμε ε, πλήρη ε, σχεδιασμό και θα πρέπει να έχουμε και βιώσιμη χρήση και ταυτόχρονα υγιές οικοσύστημα. Όπως για παράδειγμα ε, στο MSFD, στο MSFD ε, αναφέρεται σαφέστατα ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός ε, σχεδιασμός είναι το βασικό εργαλείο για να επιτύχουμε ε, συγκεκριμένους στόχους. Και μόνο μέσω βιώσιμης αλληλείας θα μπορούμε να έχουμε και βιώσιμα χωροταξικά σχέδια για τη θάλασσα, γιατί πρέπει να στηρίξουμε και τους τρεις πυλώνες που αναφέραμε σήμερα το πρωί συμμετοχή και της αλληλείας στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ε, θα είναι πιο σημαντική γιατί όπως σας είπα δεν σταματάει η αλληλεία στα χωρικά μας ύδατα. Θα πρέπει ε, να λαμβάνουμε υπόψη και το γεγονός ότι ε, τα ψάρια μετακινούνται και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το συμπεριλάβουμε και αυτό στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Okay, thank you very much, Vanessa. Um, before we go, on the προχωρήσουμε με το δεύτερο μιλτή, μήπως ε, κάνουμε ερωταπαντήσεις. Ωραία, μετά τους δύο πρώτους λοιπόν οι ερωτήσεις, θα την κρατήσω και εγώ τη δική μου ερώτηση για αργότερα. Ο λόγος στο δεύτερο μιλητή, τον David Goldsboro. Καταφθάνει. Θα μας μιλήσει για το Ολλανδικό παράδειγμα. Παρακαλώ. Okay, Καταρχήν να ευχαριστήσω τους οργανωτές για την πρόσκληση που μου απίφθηναν. Θα μιλήσω για την, ε, το χωροταξικό σχεδιασμό, διαμεθοριακό χωροταξικό σχεδιασμό στο Dogger Bank, στον αμοσύρτη του Dogger Bank. Το κεντρικό θέμα είναι οι διατρήσεις φύσεις μαζί με παράλληλα με τις αληφτικές ε, ε, δραστηριότητες. Ε, νομικό πλαίσιο, η Natura 2000 και η οδηγία για τα για το, για το θαλάσσιο περιβάλλον η u Habitat ή τα 1110 επίσης έχουμε τις νομικές υποχρεώσεις των κρατών μελών αλλά και την παράλληλη ανάπτυξη υπερολικών πάρκων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν, ε, μάλλον το, Docker Bank, ο, ο του Docker Bank ήταν ένα πραγματικό πείραμα, ε, μια μελέτη μάλλον, ε, τα, που έλαβε χώρα τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε αυτή η μελέτη με το project ε, MASPNOS, είναι μια δράση προετοιμασίας ε, χωροταξικού σχεδιασμού. Ε, συμμετείχαν η Ολλανδία, το Βέλγιο, το Ανώνα Βασίλειο και η Γερμανία. Χρηματοδοτήθηκε από το DG Mare κατά την περίοδο 2010-2012. Στόχος ήταν να διευκολύνουμε την διαμεθοριακή συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών για ένα χωροταξικό συνδυασμό που θα βασίζεται στην αρχή του οικοσυστήματος. Μετά έχουμε το Project MESMA για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των περιοχών που υπόκειται σε χωροταξικό σχεδιασμό. Ε, λίγη φέτος, ε, είναι μεγαλύτερο project με 21 εταίρους από 13 χώρες. Το, το μεγαλύτερο κομμάτι του αφιερώθηκε στο Docker Bank ε, όπου γίνεται προσπάθεια αξιολόγησης της διαδικασίας διασυνορικής συνεργασίας και συντονισμού. Να δούμε γιατί μιλάμε. Είναι ο μεγαλύτερος αμμοσύρτης της Βόρειας Θάλασσας, ε, είναι επίπεδο στη μέση, ε, ρηχός, δυναμική, δυναμικό προφίλ, καλύπτει παραπάνω από 17.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κοντινότερη γη είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, πολλά θρεπτικά συστατικά από τα οποία τα φέρνουν τα ρεύματα. Σημαντικό αλευτικό, σημαντική αλευτική περιοχή για, και, για τα αλευτικά σκάφη και περιοχή ανάπτυξης ε, ολικών πάρκων του Ηνωμένου Βασιλείου. Δανία, Ολλανδία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο ε, είναι οι γειτονικέ χώρε. Τρει χώρε, από αυτέ Γερμανία, κάτω χώρε και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν κηρύξει τμήματα του Ντάγκερ Μπάνκ ω ειδική περιοχή συντήρησης. Κάθε χώρα όμως έχει ε, τους δικούς της στόχους ΣΑΚ. ΣΑΚ είναι ειδική περιοχή ε, συντήρησης. Η Γερμανία ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, ακολούθησαν οι κάτω χώρες και τέλος το Ηνωμένο Βασίλειο. Με κάθε χώρα με τους δικούς της στόχους για το δικό τους κομμάτι, για το δικό της κομμάτι κάθε μία του Dogger Τι προσπαθούμε να προστατεύσουμε. Έχουμε πέντε ε, δεθικές κοινότητες και παρόλο ότι αυτός ο χάρτης δεν είναι πολύ λεπτομερής, είναι ε, α, αυτός πιο πολύ έχει χρησιμοποιηθεί. Δεν χρησιμοποιούμε πάρα πολύ λεπτομερείς πληροφορίες. Ε, αυτός, ο, αυ, αυτός ο χάρτης που βλέπετε είναι ο βασικός χάρτης προστασίας του Docker Bank. Στην διατήρηση αυτών των μεθικών κοινοτήτων ψαριών ε, είδαμε ότι η αλία είναι βασικό, βασική δραστηριότητα που πρέπει να ε, ε, ε, καθορίσουμε το πώς γίνεται, πού γίνεται, πρέπει να ξέρουμε πού, γίνεται, πού αλλιεύουμε, τι αλλιεύουμε και πόσο αλλιεύουμε πριν πάρουμε μέτρα. Ε, η προηγούμενη μιλήτρια έδειξε χάρτες για τη γερμανική, από τη γερμανική πλευρά. Εγώ έχω συμπεριλάβει εδώ μερικούς μικρούς χάρτες που δείχνουν ε, τις δραστηριότητε δραστηριότητες για συγκεκριμένα, συγκεκριμένους αληφτικούς στόχους, ε, στόλους συγγνώμη, και για συγκεκριμένες περιόδους. Έχουμε πολύ περισσότερα δεδομένα και αν θέλουμε να μιλήσουμε για διασυνοριακή διαχείριση θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να τα συνδυάσουμε, να τα έχουμε μπροστά μας καταρχήν και να τα συνδυάσουμε. Το 2011 μόλις αποκτήσαμε αυτά τα στοιχεία ε, η ΆΙΣΕ συζήτησε από όλα τα κράτη-μέλη να δώσουν τα στοιχεία που είχαν και αυτά τα στοιχεία που έφτασαν μας έδωσαν μια πρώτη εικόνα ε, της, ε, των δραστηριοτήτων στη νότια βόρεια θάλασσα. Εδώ έχουμε ε, την περίοδο 2007-2009, τα στοιχεία τα οποία μας δόθηκαν για αυτή την περίοδο μόνο. Ε, μιλούμε για τις δοκότρατες και τη χρήση τους σε αυτή την περιφέρεια και την συνολική ε, ένταση σε κιλοβάτ σε τη συνολική ισχύ βλέπετε ότι ε, σε, κάποια κομμάτια έχουμε ψηλή ε, ένταση, σε άλλα στα περισσότερα χαμηλότερη. Το Αρμένο Βασίλειο καθόρισε ως ένα μεγάλο κομμάτι του δικού της Docker Bank ως ΣΑΚ, ως ειδική ε, ζώνη συντήρησης. Ε, 9 γιγαβάτ θα είναι η παραγωγή του αεολικού πάρκου που χτίζει αυτή τη στιγμή ε, και θα πρέπει να το συνδυάσει με τους, ε, το Ενωμένο Βασίλειο με τους στόχους συντήρησης. Θέλω να σας πω δύο λόγια για την διαδικασία που ακολουθήθηκε όμως και θέματα διακυβέρνησης. Όλα ξεκίνησαν με το project FIMPAS. Είναι αλευτικά μέτρα σε προστατευόμενες περιοχές. Το ξεκίνησαν οι Ολλανδικές αρχές, οργάνωσαν διεθνή εργαστήρια το τρίτο από αυτά, τον Ιανουάριο του 2011, ήταν ένα διεθνέ εργαστήριο στο οποίο αναγνώρισαν ότι αν θέλουν να ασχοληθούν με το δικό τη κομμάτι του Docker Bank, δεν έχει νόημα να το κάνουν από μόνες, από μόνη από του. Πρέπει να εμπλέξουν και τα υπόλοιπα κομμάτια του Docker Bank. Γιατί, γιατί στο θαλάσσιο περιβάλλον όλα είναι δυναμικά, όλα κινούνται. Οπότε χρειαζόταν μια ομάδα, διαχειριστική ομάδα, μια διευθυντική ομάδα, steering group, ε, διασυνοριακή, δημιουργήθηκε. Είναι η Bank Steering Group, ε, η οποία δημιούργησε ένα, ε, μάλλον ζήτησε από το ΡΑΚ της Βορειάς Θάλασσας, πρόταση για την διαχείριση της αλίας ε, στην περιοχή τον ΣΑΚ του Dogger Το Steering Group απαρτίζονταν από εκπροσώπους ε, της Δανίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ISIS και βέβαια των τριών χωρών Γερμανία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν ΣΑΚ. Το ΡΑΚ της Βόρειας Θάλασσας, μάλλον το γνωρίζετε πολύ καλά, ε, ε, τα ΡΑΚ αποτελούν τμήμα τη κοινή αλληλευτική πολιτική, κατά ένα τρίτο απαραίτητο από μη κυβερνητικέ οργανώσει, από δύο τρίτα ε, το εκπροσώπου του, τομείς, του τομέα, του αλληλευτικού τομέα. Ε, το Must ε, διευκόλυνε και υποστήριξε το ράκ της Βόρειας Θάλασσας και εδώ βλέπουμε μια γραφική παράσταση, ένα χάρτη των φορέων που εμπλέκονται. Ε, το steering group απευθύνθηκε στο ράκ της Βορειας Θάλασσας, δημιουργήθηκε εκεί μια ομάδα εργασίας ε, που λειτουργήσε για, μια, για ένα χρόνο ε, με μέλη από τη Forwind, από το Maspnose, από τον ελεκτικό τομέα και από μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γι' αυτό, αλλά να σας πω ότι η εργασία, η διαδικασία ήταν πολύ εντατική, διήρκεσε πάνω από ένα χρόνο, οργανώθηκαν αρκετά εργαστήρια, αρκετά σεμινάρια, προσπαθήσαμε να δουλέψουμε μαζί για να αξιοποιήσουμε τα στοιχεία και η λειτουργία της ε, ε της Steering Group εξακολουθεί παρόλο που βρίσκεται στο τέλος της. Ε, ε, θα σας πω περισσότερο, θα εστιαστώ περισσότερο στην περίοδο 2011, Μάιος 2011 με Οκτώβριο 2011, αλλά θα σας μιλήσω και για τις σημερινέ εργασίες. Τι κάναμε, διοργανώσαμε συνεδριάσεις, χρησιμοποίησαμε ε, ε, μεγάλα διαδραστικά εργαλεία, ηλεκτρονικούς πίνακες και με, όπου χάρτες ηλεκτρονικοί, πάνω στους οποίους τοποθετούσαμε τα στοιχεία μας. ο βασικός στόχος ήταν να να αποκτήσουμε καλύτερη γνώση της κατάστασης. Οι εμπειρογνώμονες είχαν τα δικά τους λάπτοπ και γινόταν πραγματική ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις μη κυβερνικές οργανώσεις, καλής και τους προσκαλεσμένους επιστήμονες για να δούμε τι γνωρίζουμε για τον Docker Bank, τι θέλουμε να προστατέψουμε και ποιες είναι οι ενδιαφέρουσες για τους αλείς ζώνες. Επίσης είχαμε αυτό που ονομάζουμε Science on Demand, ε, δηλαδή ε, δεν καλέσαμε τους επιστήμονες να πούν στους αλλοίς τι σημαίνει στο Dogger Bank, απλώς απαντούσαν ερωτήσεις. Για παράδειγμα, στην περίοδο 2007-2009, ε, που αλλιευόταν ε, χέλη από τους Δανούς. Εκεί οι επιστήμονες δείχναν τους χάρτες και ο χάρτης είναι ενδιαφέρον γιατί το ενδιαφέρον των δανών δείχνει αυτό ο ότι δεν είναι στο επίπεδο πάνω τμήμα του αμοσύρτη αλλά στις πλαγιές του. Για ένα χρόνο λοιπόν συνεργαστήκαμε για να ε, καταλήξουμε στο αποτέλεσμα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ε, δύο ε, έγγραφα του ΡΑΚ της Βόρειας Θάλασσας που δημοσιεύθηκαν, εγκρίθηκαν από το ΡΑΚ ε, και περιλαμβάνουν ε, ένα σχέδιο διαχείρισης αλίας ε, για όλη την περιοχή που καλύπτεται από τα, από από τα τρία Natura 2000 αλλά δεν συμφωνήθηκε στον χωρισμό σε περιοχές. Γιατί τελικά οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και οι ενδιαφερόμενοι φορεί δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε ένα τελικό χωρισμό, καθορισμό ζωνών. Όμως Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του 2011, ε, το ΡΑΚ της Βόρειας Θάλασσας έγινε ε, παρατηρητής, έλαβε ε, θέση παρατηρητή στην Bank, στο, στη steering group της Dogger Bank, που στην αρχή δεν ήταν. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Εδώ έχουμε δύο χάρτες του τελικού εγγράφου. Αριστερά είναι ο χάρτης των μη κυβερνητικών οργανώσεων, δεξιά είναι ο χάρτης των αλλιέων αν ε, αναλύξετε προσεκτικά τους χάρτες θα δείτε ότι ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους. Είναι πολύ μικρές διαφορές. Ε, δεν κατάφεραν βέβαια να συμφωνήσουν τελικά, αλλά ε, συζήτησαν για το ποιες είναι οι σημαντικές περιοχές που πρέπει να απαγορεύσουμε την αλία, που πρέπει να απαγορεύσουμε άλλες δραστηριότητε κλπ. Ήταν πολύ καρποφόρα αυτή η διαδικασία. Τι έμαθα εγώ από αυτή τη διαδικασία του ράκ της Βόρειας Θάλασσας. Ήταν σημαντικό ότι καταρχήν συμφωνήσαμε για τους κανόνες του παιχνιδιού. Και με τρόπο αυστηρό. Επίσης ήταν σαφές από την αρχή, γραπτός, ε, ήταν σαφές ποιοι ήταν οι κανόνες, ε, οι ρόλοι, τα καθήκοντα του καθενός, ποια εργαστήρια θα ε, διοργανώνονταν και ποιο θα έπρεπε να είναι το παραδοτέο. Επίσης, διαφάνεια. Όλα ήταν διαφανή, κανένας δεν κρατούσε ε, κρυφούς τους στόχους του. Επίσης, ήταν πολύ σημαντικό ότι το ΡΑΚ της Βόρειας Θάλασσας διεύθυνε την διαδικασία και ε, είχε τον έλεγχό της. Ε, επίσης ήταν πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη, αμοιβαία εμπιστοσύνη και χρειάστηκε κάποιος χρόνος για να κερδιθεί αυτή. Όμω τελικά επιτεύχθηκε. Μη κυβερνητικέ οργανώσει και αλλοί εμπιστευόντουσαν ένα στον άλλο. Η... Τα μέλη του, ε, της ε, ομάδας ανέλαβαν την ευθύνη, ξεκίνησαν διάλογο βασισμένοι στο περιεχόμενο που, θέλα, που ήθελαν και στους στόχους. Τώρα, να δούμε τι λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στο Dogger Bank. Να δούμε τι μάθαμε από το χωροταξικό σχεδιασμό της θάλασσας. Ε, χρειάζονται, από την αρχή ε, διασυνορικές διαδικασίες και οι διαδικασίες θα πρέπει να, να περιγράφονται λεπτομερώς γραπτός από την αρχή. Δεύτερον, χρειάζεται να εξασφαλίσουμε διαφάνεια στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Τι σημαίνει αυτό. Πως τον έξω κόσμο χρειάζεται να είμαστε διαφανείς για το τι συμβαίνει. Για παράδειγμα, η διαδικασία του Docker Bank αυτή τη στιγμή, αν το δείτε στο ίντερνετ, θα δείτε λίγες πληροφορίες. Και αυτό είναι κρίμα. Θα έπρεπε να είμαστε σαφείς προς τον έξω κόσμο για το ποιοι είναι οι στόχοι μας. Δεύτερον, χρειάζεται διαφάνεια στο παρασκήνιο. Δηλαδή, όταν μια ομάδα ανθρώπων εργάζονται για το χωροταξικό σχεδιασμό μιας περιοχής, πρέπει να είναι ανοιχτή και διαφανής για ό,τι λάμβανε η χώρα, θα πρέπει να μοιράζονται τα δεδομένα τους ε, μεταξύ τους και μέχρι ό,τι επιτευχθεί το αποτέλεσμα να μην γίνονται διαρροές. Τέλος, θα πρέπει όλοι να ε, είναι προσιλωμένοι σε ψηλό επίπεδο. Σε χαμηλό επίπεδο είναι, ε, υπάρχει δέσμευση για συνεργασία με τους γείτονες, αλλά σε υψηλότερο επίπεδο έχουμε τη διαβούλευση η διαβούλευση δεν σημαίνει απλώς ε, ρωτάω και δίνω απαντήσεις. Είπα, έχει μια πιο σημαντική δέσμευση και σε ακόμα πιο ψηλό επίπεδο υπάρχει συντονισμός. αυτό είναι το ψηλότερο επίπεδο δέσμευσης και προσήλωσης. Ο χωροταξικός σχεδιασμός ε, μπορεί και πρέπει να αποφελθεί από τη χρήση γεωχωρικών ε, εργαλείων. Γιατί μας ε, βοηθούν να δούμε τι στοιχεία έχουμε και τι στοιχεία μας λείπουν. Άλλα σημαντικά στοιχεία είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη εντολή. Άνθρωποι οι οποίοι συζητούν γύρω από ένα τραπέζι στο χωροταξικό σχεδιασμό πρέπει να έχουν μια εντολή. Και σε αυτή τη διαδικασία του Dogger Bank η εντολή δεν ήταν σαφής. Δεν ήταν σαφές ποιος έχει εντολή, οι αρχές ή οι εμπλεκόμενοι φορείς. Γιατί το να μιλάει κανείς για χωροταξικό σχεδιασμό χωρίς εντολή δημιουργείται πρόβλημα. Δημιουργεί πρόβλημα. Μετά, η χρηματοδότηση της συμμετοχής των ε, εμπλεκομένων. Ε, χρειάζεται να αφιερωθεί πολύς χρόνος ε, και συνεπώς αυτό έχει κόστος. Αν δεν είχαμε τη χρηματοδότηση της Mare, δεν θα μπορούσε να έχει λάβει χώρα αυτή η διαδικασία. Και τέλος θα πρέπει να ακολουθείτε η προσαρμόσιμη διαχείριση. Δηλαδή έχουμε λίγα πράγματα, ε, έχουμε λίγες γνώσεις για τις επιπτώσεις της, των ελευτικών δραστηριοτήτων. Πρέπει λοιπόν να ε, ε, εντοπίζουμε, να παρακολουθούμε το πώς η διαχείριση, τις επιπτώσεις διαχείρισης και να την προσαρμόσουμε. Τέλος, ποιος είναι ο ρόλος των επιστημόνων. Προφανώς το πείραμα αυτό ήταν επιστημονικό, πείραμα επιστημονική μελέτη, συνεπώς χρησιμοποίησαν πολύ τους επιστήμονες, ε, η ISIS ε, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο γιατί, κυρίως γιατί το, Υπουργό, το ε, Ολλανδικό Υπουργείο Οικονομικών έχει στενές σχέσεις με την ISIS. Αυτό αποτελεί περιορισμό γιατί κάποια πράγματα είχαν ήδη συμφωνηθεί. Αν δούμε όμως το τι συμβαίνει με το ρόλο της επιστήμης, γενικά είναι, χα... είναι μικρός, δευτερεύον. το steering group της, του Docker Bank είχε συμφωνήσει να χρησιμοποιήσει ένα περιορισμένο ε, όγκο δεδομένων και αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν όλα τα δεδομένα ούτε και αξιολογήθηκαν όλα τα σενάρια. Αυτό δυσχεραίνει την πρόβλεψη των επιπτώσεων των μέτρων που μπορούν να ληφθούν. Η συμφωνία να χρησιμοποιηθεί ένα συγκεκριμένο dataset ε, δημιούργησε πρόβλημα και στην διεύρυνση της βάσης δεδομένων. Αυτό, συμφωνούν οι περισσότεροι, είναι σημαντικό εμπόδιο ε, για τον Bank, αλλά και αλλού. Πρέπει να μπορέσουμε να διευρύνουμε τη γνώση μας. Μετά, οι, αυτοί που, αποφασίζουν από, που λαμβάνουν τις αποφάσεις ε, πρέπει να συνεργάζονται επικοδομητικά με τους επιστήμονες. Αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Ε, εμείς είδαμε το διάλογο για, να λαμβάνει χώρα για το περιεχόμενο, ε, αλλά μετακινηθήκαμε από το διάλογο σε διαπραγμάτευση και στην διαδικασία του Dogger Bank, η διαδικασία του Dogger Bank ήταν πιο πολύ μια διαδικασία διαπραγμάτευση τελικά και όχι διαδικασία αμοιβαία ε, διεύρυνση των γνώσεων. Και αυτό είναι κρίμα. Θα έπρεπε να μιλήσουμε για το περιεχόμενο, για τις, το, για τις και τα δεδομένα πιο πολύ. Αυτά είχα να πω σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που μου δόθηκε. Αυτή είναι η εμπειρία μας για το αμοσύρτη του Dogger Bank. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να ληφθούν όλα αυτά υπόψη στην ε, διατύπωση της νέας οδηγίας. Ευχαριστώ πολύ, Ντέιβιτ. Ακούσαμε τους δύο μιλητές μας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Είδαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχουν όλες οι ενδιαφερόμενες μονάδες ήδη από την αρχή της διαδικασίας, αλλιώς δεν θα πετύχουμε μια καλή λύση. Είδαμε τι συγκρούσεις υπάρχουν ανάμεσα στις, στα αιωλικά πάρκα, την Αλία κλπ. Ο Ντέιβιντ δεν φαίνεται απόλυτα ικανοποιημένο με τα όσα συμβαίνουν. Ε, σίγουρα υπάρχει ε, περιθώριο βελτίωση. Ε, Πρώτα να δώσω το λόγο στου άλλου. Μία ερώτηση προ τη Βανέσα. Κάτι που δεν ανέφερε και που εμένα πάντα με ενδιαφέρει. Είναι τα αιωλικά πάρκα και η ηχθειοκαλλιέργεια και ο συνδυασμό του. Μπορεί να μην είναι το, η λύση για όλα, αλλά μήπω μπορεί να αναφερθεί στο θέμα αυτό. Ναι. Ε, ιδιαίτερα το Ινστιτούτο Αλφαβέγγλης στην Γερμανία σκέφτεται πώς μπορεί να ε, ενσωματώσει τις, ε, την ηχθειοκαλλιέργεια στα θαλάσσια ολικά πάρκα. Έχουν γίνει έρευνες. Υπάρχουν λοιπόν ήδη τεχνικές λύσεις, αλλά επειδή μιλάμε για θαλάσσια ολικά πάρκα, αν αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές. Πάντως πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε σχετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως σας είπα δεν είναι ε, λύση για όλα αυτά. Τα ψάρια θα πρέπει να κολυμπάνε ελεύθερα, όπως πάντα έκαναν, ε, αλλά καθότι χρειαζόμαστε περισσότερα ψάρια στο μέλλον από ό,τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, ε, ίσως θα ήταν χρήσιμο ένας χώρος να χρησιμοποιείται για δύο δραστηριότητες. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους άλλους συμμετέχοντες να θέσουν ερωτήσεις ή να κάνουν παρατηρήσεις. Ιζαμπέλα, παρακαλώ. Merci beaucoup, merci. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους ομιλητές μας που με τα παραδείγματά τους αυτά διευκρίνησαν περισσότερο και εμβάθυναν με πολύ πιο ενδιαφέροντα τρόπο τα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ιδίω πρέπει να πω ένα πρόβλημα το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά την άποψή μου, ίσως θα πρέπει να το επεξεργαστούμε και αυτό, και αυτό είναι το θέμα τη διακυβέρνηση. Διότι βλέπουμε και στα δύο παραδείγματα ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα συνεργασία, διαβούλευση, όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε κατά νου και ως πρώτη αντίδραση νομίζω θα έλεγα ότι θα πρέπει να έχουμε συνεργασία στη διάρκεια των εργασιών και ε, διαβούλευση κατά την επαλήθευση, αλλά θα πρέπει να τα συζητήσουμε βέβαια όλα αυτά, αλλά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ε, όλοι όσοι μίλησαν όμως σήμερα το πρωί μας είπαν ότι ότι οι συζητήσεις πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με τους ενδιαφερομένους και όχι μόνο κατά τη στιγμή της λήψης της απόφασης, γιατί ε, σε αυτή την περίπτωση βρισκόμαστε ενώπιον της αποτυχίας. Και υπάρχει και μία συζήτηση ε, την οποία ξεκίνησε ο κύριος Γκένσπορο. Νομίζω ότι είπατε, αλλά δεν κατάλαβα απολύτως, ότι η διατησία πιο πολύ ήταν υπομορφή διαπραγμάτευσης και όχι ε, εκπόνησης ενός προγράμματος. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο παράδειγμα το αναφέρατε συγκεκριμένα. Και εγώ είχα μια άλλη εμπειρία για ε, την περίπτωση της Βρετάνης, στην οποία αναφέρθηκε ο συνάδελφος Πιέρν Καρνετσκίν και σε χωροταξικό σχεδιασμό, όπου καταλήξαμε τελικά σε συμβιβασμό. Δηλαδή, υπήρχε μία περιοχή παράκτιων ολικών ε, πάρκων ε, που χρηματοδοτούσαν ε, οι βιομηχανίες ενέργειας, διότι βρισκόταν σε μία περιοχή που ήταν αρκετά ευαίσθητη ώστε να μπορέσει, ώστε τελικώς προκειμένου να μπορέσει να κατασκευαστεί, ε, ήταν ιδιαίτερα δαπανερή. Αυτό είχαν επιλέξει, αλλά ε, όπως είπε και ο συνάδελφος, ήταν στην περιοχή καλλιέργειας ε, των χτενιών. Και τι γίνεται, ξεκίνησε μια ολόκληρη συζήτηση και μετά από ε, μελέτη επιπτώσεων κοινωνικών και οικονομικών αποφασίστηκε ότι όντως ο πλούτος που παράγεται από τα χτένια είναι σημαντικός και ε, ίσως ο πλούτος ο οποίος θα προκύψει από το ελληνικό πάρκο να είναι και αυτός εξίσου σημαντικός, αλλά για να μπορέσουν να συμβιώσουν θα ε, πάει λίγο πιο βόρεια η εγκατάσταση των, ε, του ελικού πάρκου και ε, θα στοιχήσει και αυτό βέβαια λίγο ακριβότερα διότι θα υπάρχουν περισσότερα καλώδια γιατί ε, θα είναι πιο σημαντικά τα θεμέλια και το καθεξής αλλά τελικός ο συμβιβασμός στο οποίο καταλήξαμε ήταν κέρδος για τις ενεργειακές επιχειρήσεις διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πιο ασφαλείς επενδύσεις Υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες είναι και πιο νομικά ε, ασφαλείς και γνωρίζουμε ότι δεν θα υπάρξει και πρόβλημα συνύπαρξης τουλάχιστον ε, για τα χτένια. Δεν θα ε, πω περισσότερα, απλώς ήθελα να πω ότι όταν αναφερόμαστε σε συγκεκριμένε εντολές και συμφωνώ πολύ αυτό που είπατε ότι θα πρέπει να τεθεί και το ζήτημα της εντολής, θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι θέλουμε. Τι θέλουμε, κατά την άποψή μου, ένα συμβιβασμό. Προφανώς και ένα συμβιβασμό. Ε, ο συμβιβασμός όμως που περνά ε, από μία διαπραγμάτευση που είναι περίπου ότι ε, αν δεν δεχτείτε αυτό που σας λέμε θα σας τραβήξουν το χαλί κατά τα πόδια δεν είναι σωστός. Χρειάζεται ένας συμβιβασμός στον οποίο θα υπάρχουν συγκεκριμένε παράμετροι. Δεν θα βρούμε εδώ ποιες θα είναι αυτές οι παράμετροι. Ε, ε, και θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν τελικώς ε, τι σας δίδαξε αυτή η διαπραγμάτευση και μετά αναφερθήκατε και εσείς στο θέμα της διακυβέρνησης, την ανέφεραν και διάφοροι άλλοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει συζήτηση, συνεργασία κατά τη διάρκεια της εκπόνησης ε, οποιοδήποτε έργο και τελικώς ε, τελική διαβούλευση με όλους όσους ενδιαφέρονται για το θέμα. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Δεν ήταν ερώτηση. David, όμως, θέλετε να σχολιάσετε. Θα πω κι εγώ κάποια πράγματα για τη διακυβέρνηση στη συνέχεια. Ναι, θα ήθελα να σχολιάσω. Νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ε, αυτή η διαδικασία στο Dogger Bank ξεκίνησε χωρίς ε, τίποτα υπήρχε ένα αίτημα από την Περιφερειακή Οργάνωση της Βόρειας Θάλησης και αυτοί είχαν μια ολόκληρη διαδικασία, τα πάντα ήταν γραμμένα και η υπόθεσή τους ήταν ότι θα υπήρχε η ίδια δομή και η ίδια διαδικασία που θα βοηθούσε την όλη διαδικασία. η αποστολή ε, των κρατών μελών ε, προς το περιφερειακό ΡΑΚ ήταν να τους κάνουν μια πρόταση και τελικώς δεν ήταν καλό γιατί ε, τους επιβάρυναν με κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να λύσουν. Θα μπορούσαν να κάνουν προτάσεις αλλά η απόφαση έπρεπε να είναι στα χέρια αυτών που χαράσουν την πολιτική και αυτό θα έπρεπε να είχε υποθεί ευθύ εξ αρχής θα γίνουν προτάσεις από το ε, Περιφερειακή Οργάνωση της Βόρειας Θάλασσας και θα αποφασίσουν οι ηθήνοντες. Και θα είχε τελειώσει και το ζήτημα και δεν θα είχε δημιουργηθεί το θέμα με το ε, Περιφερειακή Οργάνωση της Βόρειας Θάλασσας. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο λοιπόν ποιο έχει καθήκον να κάνει τι. Και συμφωνώ και μαζί σας ότι αυτό πρέπει να γίνεται ευθύ εξ αρχής. Ε, και εάν από εκεί και πέρα οι αρχές υποχρεωθούν να έχουν διαδικασίες, να γράφουν ποιος θα αποφασίσει, πότε θα το αποφασίσει, επί τη βάση ποιου πράγματος, τότε τα πράγματα θα είναι σαφέστερα και η όλη διαδικασία θα είναι καλύτερη. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ωραία, ευχαριστώ, Ντέιβιτ. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι κι εγώ. Η Ζαμπέλ πολύ σωστά είπε ότι δεν υπάρχει κατάλληλη διακυβέρνηση στην πρόταση για τον ε, θαλάσσιο χωροταξικό ε, σχεδιασμό δεν υπάρχει άρθρο που να λέει ότι η διακυβέρνηση είναι σημαντική, αλλά η διακυβέρνηση διέπει ουσιαστικά όλα τα άρθρα, διότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε ε, διπλές εργασίες, καλύτερες λύσεις, να μην υπάρχει τόση γραφειοκρατία και φυσικά η διακυβέρνηση είναι υψίστης της σημασίας για όλη τη διαδικασία του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Ένα-δυο λεπτά, ε, ε, ο κύριος Πρόεδρος. Το άλλο θέμα που κατάλαβα από όλες τις συζητήσεις σήμερα το πρωί είναι είναι ο αντίκτυπος ε, των ε, θαλάσσιων ολικών πάρκων. Ε, οι εταιρείε ενέργειας επιλέγουν αβαθή ύδατα κοντά στην ε, στεριά επειδή είναι πιο φτηνή η κατασκευή, είναι πιο εύκολο να ε, βάλει κανείς καλώδια. Ε, αυτά όμως είναι καλύτερα μέρη για ψάρεμα. Χαίρομαι λοιπόν που καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια να λυθούν οι διαφορές αυτές. Κανείς δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι η αιωλική ενέργεια μάλλον είναι ο πιο ακριβώς και άχρηστος τρόπος παραγωγής ενέργειας ε, για την ανθρωπότητα. Μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε τα ερήπια αυτών των τερατουργημάτων ε, να καταστρέφουν τα τοπία μας ε, και την ύπεθρό μα ε, Στο Humberside στην Αγγλία, στην ακτή, η Dong Energy της Δανία εταιρεία ε, κατασκευάζει τεράστιο ολικό πάρκο το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ε, τα καβούρια και τις καραβίδες εκεί. Και οι αλληλείς που πάντα ψάρευαν εκεί θα χρειάζονται άδεια από την Dong Energy για να πλησιάσουν ε, περισσότερο από 500 μέτρα ε, τις ε, τουρμπίνες αυτές, τους Ε, Ξαφνικά λοιπόν οι αλληλείς που επί χρόνια αλλιεύουν εκεί πέρα πρέπει να πάρουν τηλέφωνο μια ξένη εταιρεία για να πάρουν άδεια σε να αλλιεύουν εκεί που πάντα ψάρευαν. Ε, εάν δεν μπορέσουμε να λύσουμε τέτοια προβλήματα, τότε ήταν ε, ε, μάταιη η συζήτηση που είχαμε σήμερα. Αυτά τα προβλήματα θέλουμε να λύσει η οδηγία αυτή. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είδαμε ότι υπάρχουν τρόποι να λυθούν τα προβλήματα αυτά, αλλά ελπίζω να μην είναι όλα μάταια επειδή η όλη η ιστορία με τους ανεμόμυλους κατά τη γνώμη μου είναι τελείως άχρηστη και βασίζεται στις επιδοτήσεις. Ε, κύριε Μάισνερ, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα συζητήσουμε αυτό. Η Ισαπέλ για μια σύντομη παρατήρηση και μετά έχουμε άλλη μια ερώτηση. Θα ήθελα να προσθέσω το εξή. Συμφωνώ με τα όσα είπε και ο Στίβενσον. Να προσθέσω το εξή όμω. Χωρί προγραμματισμό θα είναι Δαβίθ εναντίον Γολιάθ. Και ο πιο δυνατός θα κερδίσει. Χωρίς αυτό να αποτελεί να είναι υπέρ του γενικού συμφέροντος. Συνεπώς ο σχεδιασμός θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα των προσανατολισμών μας γιατί ο σχεδιασμός μπορεί να έχει και πρέπει να έχει ως στόχο το συνολικό γενικό συμφέρον. Θα λαμβάνει υπόψη κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, καθώς επίσης και την ισορροπία μεταξύ τους, προκειμένου να αποφύγουμε το δίκαιο του χειροτέρου. Okay, thank you, Isabel, for Ωραία, ευχαριστούμε, Ιζαμπέλ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο εξώ από την κυρία εκεί. Δύο. Εσάς τους δύο και μετά θα πρέπει να κλείσουμε. Καλή σας μέρα. Ε, δουλεύω για την ε, βιομηχανία ολικών ε, πάρκων στη θάλασσα. Δεν θα μπω συζήτηση αν είναι κάτι καλό ή όχι. Ε, σε ε, στιγμή κρίσης είναι καλό να αναπτύσσονται δραστηριότητες στη θάλασσα, κάτι που θα μπορούσε να μας οδηγήσει να βγούμε από την κρίση. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Ε, η... Έχουμε μιλήσει για διαβούλευση και η... εμείς θέλουμε να διαβουλευτούμε με όλους τους υπόλοιπους τομείς. Για παράδειγμα στο Σεμπριέ, το οποίο προβλήθηκε ως παράδειγμα και πολύ σωστά, είναι ένα παράδειγμα ε, ε, που προχωρήσαμε πολύ γρήγορα χάρη σε αυτή τη διαβούλευση που έγινε. Και εμείς έχουμε υποχρεώσεις και οι άλλοι έχουν υποχρεώσεις. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι, σε σχέση με αυτήν την οδηγία, είναι ότι ε, σε συνεργασία έχουμε μιλήσει και με μη κυβερνητικέ οργανώσει όπως τη ΒΒΕΦ και ε, χαιρόμαστε που θα υποβληθεί αυτή η νομοθεσία διότι θα δίδει ένα ορισμό του χωροταξικού σχεδιασμού στη θάλασσα για όλα τα κράτη-μέλη, κοινό. Και μετά το κάθε κράτο μέλο θα πρέπει να προβεί σε αυτό το σχεδιασμό. Και μέσω αυτού μπορεί να δοθεί η ευελιξία που χρειάζεται ε, και ο αληθικό τομέα και εμεί. Και σίγουρα το ονομαστικό κείμενο θα προβλέπει και την υποχρέωση διασυνορική συνεργασία. Εμεί ζητούμε από το Κοινοβούλιο να είναι φιλόδοξο ω προ τι απαιτήσει του. Οι διαπραγματεύσει λαμβάνουν χώρα στο Συμβούλιο, δεν είναι εύκολε ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προασπιστεί την ε, σύνδεση ανάμεσα στην στεριά και τη θάλασσα και να υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν το χρονοταξικό του σχεδιασμό με βάση ένα συγκεκριμένο όραμα. Χρειαζόμαστε στόχους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τέλος, ζητούμε από τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη και τις ανανεώσιμες στη θάλασσα και τις αλληλευτικές δραστηριότητε. Ε, πιστεύουμε πολύ στο ρόλο του Κοινοβουλίου σε αυτό. Well, uh, uh, um, uh, Ασφαλώς. Η Επιτροπή Μεταφορών σήμερα ε, ε, ψήφισε την έκθεση για τη γαλάζια ανάπτυξη η οποία θα είναι τμήμα της ε, στατικής Ευρώπης 2020 η γαλάζια ανάπτυξη σημαίνει περισσότερη ε, χθιοτροφία, περισσότερη αλεία, ε, ε, μπλε βιοτεχνολογία, γαλάζια βιοτεχνολογία, οι πρώτε ύλε από τη θάλασσα, όλοι αυτοί είναι τομεί που αναπτύσσονται και ασφαλώς θα πρέπει να βρούμε λύσεις που να μας βοηθούν να αποφύγουμε σύγκρουση, συγκρούσεις και να μας βοηθήσουν επίσης να αναπτύξουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες με ένα λογικό τρόπο ε, έτσι ώστε όλες αυτές οι δραστηριότητες να συνυπάρχουν ειρηνικά. Και κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Good uh, morning. My name is uh, Milos. Καλημέρα, λέγομαι Μίλος Λάποβιτς, ε, εκπροσωπώ τις ε, ε, Ολλανδικές ε, παράκτιες περιφέρειες εδώ στις Βρυξέλλες. Όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμμεριζόμαστε τη φιλοδοξία ε, να αναπτυχθεί η γαλάζια οικονομία της ε, Ευρώπης ε, και να έχουμε ολοκληρωμένη διαχείριση της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών. Πιστεύουμε ότι κατευθυντήρες γραμμές για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη διαχείριση της θάλασσας έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν την βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, έχουμε κάποιες ανησυχίες διότι φοβόμαστε ότι μια τέτοια οδηγία θα οδηγήσει σε περισσότερη ευρωπαϊκή νομοθεσία εντός των συγκεκριμένων τομέων πολιτικής και αναρωτιόμασταν εάν η οδηγία είναι το κατάλληλο μέσο. στα προηγούμενα έγγραφά μας ε, θεωρήσαμε ότι, η ε, ανοιχτή μέθοδος ε, συντονισμού, θα είναι πιο κατάλληλο μέσο για να πετύχουμε το στόχο μας. Πέρα από αυτό όμως, οι πέντε αυτές περιφέρειες πιστεύουν ότι θα πρέπει οποιοδήποτε νομικό μέσο να περιορίζεται στον συντονισμό. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν χέγγια στην οδηγία ώστε ε, να μην ε, υπάρχουν ε, περισσότεροι και νέοι κανόνες για τον χωροταξικό σχεδιασμό. Καταλαβαίνετε ότι ως αυτοί που εφαρμόζουν τον χωροταξικό σχεδιασμό στις παράκτιες περιοχές πιστεύουμε ότι οι στόχοι που περιλαμβάνονται στην οδηγία και αυτοί που δεν υπάρχουν ακόμα στην οδηγία, για παράδειγμα όπως είναι η στέγαση, ε, θα υπάρξουν συγκρούσεις ανάμεσα σε αυτούς τους τομείς ε, και επίσης ε, κατά τον χωροταξικό σχεδιασμό πάντα έχουμε διαβουλεύσεις με ομάδες ενδιαφερομένων. Οι ενδιαφερόμενοι όμως, εάν ε, δεν είναι ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα ενός τέτοιου σχεδίου, θα έχουν τη δυνατότητα ε, από την οδηγία αυτή να ε, μπλοκάρουν, να σταματήσουν την ανάπτυξη σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, Κάποιοι που να μην είναι ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα των σχεδίων που θα παρουσιάσει η Επιτροπή. Θα μπορέσουν να παρεμποδίσουν ε, ε, σχέδια οικονομικής ανάπτυξης όπως είναι ο τουρισμός, ε, η στέγαση, η υποδομή κλπ. Μπορείτε παρακαλώ να κλείσετε διότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ναι, φυσικά. Τέλος, ανησυχούμε ότι το διοικητικό άχθος ε, θα αυξηθεί με την οδηγία αυτή και γι' αυτό προτείνουμε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπάρχουσες πολιτικές από τα κράτη-μέλη και διαδικασίες. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε ε, ε, δική μας πράξη για τον χωροταξικό σχεδιασμό που προβλέπει δεκαετή προθεσμία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, συζητήσαμε την οδηγία για τον ε, θαλάσσιο χωροτεξικό σχεδιασμό. Ε, η διαδικασία αυτή μόλις ξεκίνησε. Θα συνεχιστούν λοιπόν οι συζητήσεις. Εγώ θα εκπονήσω την έκθεση αυτή για το Κοινοβούλιο. Οποιοςδήποτε λοιπόν θέλει να σχολιάσει μπορεί να το, έχει, μπορεί να το, μπορεί να το κάνει. Ε, δύο ομιλητέ ακόμα έχουμε. Λείπαμε, μόλι έκλεισα τον κατάλογο των ομιλητών. Πρέπει να κλείσουμε. Δεν είναι όμω η τελευταία συζήτηση ε, για τον χωροταξικό σχεδιασμό. σω θα πρέπει η Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα να πει λίγα λόγια τώρα στο τέλο. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και Ε, Πολλά από τα παραδείγματα που μας δόθηκαν ε, δείχνουν πολύ ε, καλά ποια είναι η κατάσταση. Θα είναι χρήσιμο να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. to speak as well. So really, I think we have to close right now. She's a member of. The I know, I know. Committee. You wanted to say something as well because uh, we had to. Θέλετε κι εσείς να πείτε κάτι, διότι είχαμε άλλους δύο μιλητές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Αν είσαστε πολύ σύντομοι. Ναι, ναι, θα είμαι πολύ σύντομη. Ευχαριστώ πολύ τους συζητητές. Αλλά να σας πω ποιες είναι και οι δικές μας προσπάθειες. Πρέπει να το εκθέσουμε κι αυτό. Τρεις είμαστε μόνο παρόντες που τους ακούμε. Ε, κάτι έχουμε να πούμε κι εμείς. Να σας πω για το εξή ζήτημα. Για να σας πω για αυτό το ζήτημα ότι ήμουν εισηγήτρια από την ομάδα μου. Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται να γίνεται ισορροπημένο χωροταξικός ε, σχεδιασμός ε, χωρίς ε, σύγκρουση των δράσεων και των χρήσεων υπό την προϋπόθεση ότι προσπιζόμαστε το οικονομικό και κοινωνικό συμφέρον της αλίας, του περιβάλλοντος, αλλά εγώ είμαι υπέρ και της ενέργειας. Στην χώρα μου έχουμε διάφορα project, στην Ορμανδία επίσης ε, ε, είδα ότι αλληλείς ε, ενδιαφερόμενοι φορείς, επιχειρήσεις παροχής ενέργειας διαβουλεύθηκαν, συζήτησαν, συνεννοήθηκαν με καλά αποτελέσματα και πρέπει να κάνουμε το ίδιο διότι οι παράκτιες περιοχές έχουν να ωφεληθούν από τα πρόσβητα αυτά τα ενεργειακά στη θάλασσα. υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, να γίνουν σωστά τα πράγματα υπό την προπόθεση ότι ε, συνεργαζόμαστε όλοι οι τομείς που λειτουργούν και χρησιμοποιούν το θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ καλή η δουλειά σας. Πολύ καλή ε, πολύ καλή η δουλειά μας και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε παρόντες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την προσθήκη. Τελειώνω το πάνελ, μου δίνω το λόγο στον πρόεδρο για να κλείσει. Ευχαριστώ πολύ εσάς, την κυρία Τόμα, την κυρία Πατραουνέβες που χρειάστηκε να φύγει και όλους τους ομιλητές που πήραν μέρος. Έγινε σαφέστατο ότι υπάρχουν πολλές επικαλυπτόμενες δραστηριότητες ανεμογεννήτριες, ε, ανανεώσιμες πηγές στη θάλασσα, τουρισμό, εξορυκτική βιομηχανία, αλληλεία κλπ. κλπ. Ε, χρειάζεται μια ολοκληρωμένη διαχείριση των πράκτιων ζωνών, χρειάζεται χωροταξικό σχεδιασμό, αυτά είναι προφανή πια. Ε, ήταν πάρα πολύ επίκαιρη και κέρια η σημερινή συζήτηση. Σας ευχαριστώ όλους που λάβατε μέρος. Τούτου λεχθέντος η Επιτροπή Αλίας εξεκολουθεί να ε, συνεδριάζει. Φτάσαμε στο σημείο 19 της ημερησίας διάταξης. Έχουμε τα διάφορα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος θέλει να σχολιάσει οτιδήποτε στα διάφορα. Αν όχι, περνάω στο σημείο 20. Ανακοινώσεις του Προέδρου για τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές. Έχετε ένα έγγραφο. Η χτεσινή συνάντηση των συντονιστών διήρκεσε πολύ λίγη ώρα. Ε, κατανείμαμε κάποιες εκθέσεις μεταξύ των ομάδων. Έχετε τις αποφάσεις που ελήφθησαν ε, γραπτός. Σημείο 21, προσεχή συνεδρίαση, προσεχή συνεδρίαση 17 Ιανουαρίου και 18 Ιουνίου του 2013. Σας περιμένουμε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς και τους διεθνείς.